Να αρχίσουμε συνάδελφοι με το δεύτερο μέρος της ακρόασης για το, τη δέσμη μέτρων για τις ιδεοδομικές μεταφορές. Τώρα θα μιλήσουμε για ασφάλεια και τεχνικές προδιαγραφές. Έχουμε πέντε προσκαλεσμένους ομιλητές και μετά θα μιλήσουν οι σκιώδεις, ε, όχι, οι και μετά οι συντονιστές. Ο πρώτος ομιλητής θα μας μιλήσει για την σκοπιά των κατασκευαστών. Ο κύριος Χωσέ Κορτάζ Ομπιέτα που είναι τεχνικός διευθυντής τη CIF Μπεσάν στην Ισπανία και είναι και μέλος της UNIFE. Κύριε Ομπιέτα, έχετε το λόγο. Μην υπερβείτε το δεκάλεπτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω την σκοπιά των κατασκευαστών για την διαλειτουργικότητα που είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας και για όλους τους κατασκευαστές. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα Δύο σημαντικά πράγματα πρέπει να δούμε, τη συνθετότητα και την ε, δαπανηρότητα και το χρονοβόρο τη χρονοβόρο διαδικασία. Χρειάζονται διαφορετικές άδειες από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη επίσης εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες και εκτός από το TSI, τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, Υπάρχουν και 11.000 περίπου διαφορετικοί εθνικοί κανόνες, οπότε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και βέβαια δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Είναι και δαπανηρό και χρονοβόρο. Έχουμε υπολογίσει ότι 1,2 δις ευρώ ε, οχήματα περιμένουν την άδεια. Δηλαδή αυτά είναι χρήματα, είναι επενδεδημένα σε οχήματα και πολλές φορές οι διαδικασίες ε, αδειοδότησης υπερβαίνουν τα δύο χρόνια. Έχουμε το θέμα της ε, διαποδοχής ή της διακρατικής αποδοχής. Στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι ήταν αυτή η λύση, αλλά και πάλι έχουμε τους 11.000 ε, τεχνικούς κανόνες, οπότε είναι πολύ δύσκολο πρακτικά να ισχύσει αυτή η διαποδοχή, η διακρατική αποδοχή ο κλάδος χρειάζεται ε, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό φορέα θα είναι μία αδειοδότηση και θα είναι ενοποιημένες οι διαδικασίες και οι κανόνες γιατί τα κράτη εφαρμόζουν άλλες διαδικασίες και κανόνες. Οπότε ναι, χρειάζονται ενοποιημένες διαδικασίες και ενοποιημένοι κανόνες. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση το σημερινό σύστημα. Ξέρετε τα νόμπος και τα ντέμπος αυτούς τους φορείς κοινοποίησης και ανάθεσης. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας τεχνικός φάκελος με πάρα πολλά έντυπα που παρουσιάζουν τα διάφορα πρότυπα και αξιολογούνται από τους φορείς κοινοποίησης που βλέπουν τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και αξιολογούνται και από τα ντέμπος φορείς ανάθεσης που αξιολογούν τους εθνικούς κανόνες συνήθως. Οπότε όταν ετοιμαστεί ο τεχνικός φάκελος πάτε για εξουσιοδότηση στις διάφορες χώρες. Θα πάτε στην Εθνική Αρχή Ασφάλειας της πρώτες χώρες, της δεύτερης, της τρίτης κλπ. κλπ πριν περάσουν στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτό δε. Είναι ότι οι διαδικασίες διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Τι περιμένουμε λοιπόν εμείς. Περιμένουμε ο ΕΟΣ είναι μονοθυριδική υπηρεσία που θα ξεπεράσει τα σημερινά εμπόδια Βέβαια, ο τεχνικός φάκελος θα πρέπει να προετοιμαστεί, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί από του φορείς ανάθεση κοινοποίηση, αλλά η εξουσιοδότηση θα δίνεται από τον ΕΟΣ, που θα δρά ως μονοαπευθυντική ε, υπηρεσία και μετά θα αποφασίσουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ε, να περάσουν σε εμπορική χρήση ε, ενημερώνοντας το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και δεν μπορούμε να αλλάξουμε εννιά νυχτή τα πράγματα. Αυτό θα ήταν απολύτως αδύνατον. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι εμείς ε, μπορούμε να έχουμε ένα, ε, τον ετούντα ε, στον ΕΟΣ και μετά να περνούν στις εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες οι πληροφορίες για να παίρνουμε τα σχόλια και την αξιολόγηση συμβατότητας από τις εθνικές υπηρεσίες για να μην λησμονηθεί και ε, κάποιο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Και μετά οι εθνικές υπηρεσίες επανέρχονται στον ΕΟΣ που είναι ο Εθνικός Οργανισμός Ιδροδρόμων που θα αποφανθεί. Θα πρέπει ο ΕΟΣ λοιπόν όπως είπα να είναι απόλυτα μόνο επιθυντικός φορέας σχετικά με την έκδοση τη άδεια του οχήματο ποιος, ποιος είναι ο τομέας χρήσης που πρέπει όλοι να τηρούμε. Είναι οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ε, συνήθως ε, οι φορείς κοινοποίηση την εξετάζουν και όλοι οι εθνικοί κανόνες που είναι υποχρεωτικοί και πρέπει να συμμορφωνόμαστε προς αυτούς όλοι και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να αξιολογείται που είναι η συμβατότητα μεταξύ οχήματο και δικτύου ή των ομάδων δικτύων γιατί λειτουργούν διασυνοριακά και πάμε από το ένα δίκτυο στο άλλο και εκεί μπορεί να υπάρχει διαφορά προτύπων. Και βέβαια σε αυτή τη μεταβατική περίοδο είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο ΕΟΣ δεν μπορεί από την πρώτη μέρα να λειτουργήσει και κάποιος νομίζω σήμερα το είπε αυτό ε, όταν μιλούσε για υπεργολαβικές διαδικασίες. Η εξουσιοδότηση, η αδειοδότηση του οχήματο θα μπορέσει να δουλέψει με δύο τρόπους. Αν είναι για περισσότερο από ένα κράτο μέλος, τότε θα πρέπει να δίνεται από τον ΕΟΣ η άδεια του οχήματο. Και βέβαια θα μπορεί και η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας να τα παρακολουθεί όλα αυτά, γιατί τώρα ο ΕΟΣ δεν έχει τη δυνατότητα να καταπιαστεί με όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, θα πρέπει όταν είναι ε, η διοδότηση από ένα κράτος μέλος θα μπορεί και η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας να εξουσιοδοτεί και θα μπορεί ο ετών να επιλέγει ή από τον ΕΟΣ ή από το εθνικό επίπεδο. Σε τελευταία ανάλυση όμως ε, θα πρέπει ο τελικός στόχος να είναι, να είναι μόνο απευθυντική υπηρεσία ο ΕΟΣ σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας. Οι διαδικασίες όμως είναι πολύ σημαντικές και υπάρχουν πολλοί κανόνες. Τα είπαμε αυτό. Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικοί και πολλοί κανόνες. Παράλληλα λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε δουλειά πάνω στη δυνατότητα να, το ενδεχόμενο, να μειώσουμε άχρηστους εθνικούς κανόνες. Ε, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα τέτοια περιθώριο πολύ αυτό δε, πάλι δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε πάνω από τριετία για να τα μειώσουμε. Αυτό όμως είναι υποχρεωτικό για όλους μας. Γιατί μάλλον σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι άχρηστοι οι εθνικοί κανόνες, δεν εξυπηρετούν τίποτε. Για να τελειώσω λοιπόν Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για την, ε, το νέο σύστημα ευρωπαϊκής αδειοδότησης. Ε, θα πρέπει ο ΕΟΣ να είναι υπεύθυνο για την διαδικασία αδειοδότησης, να είναι μονοαπευθυντική, να είναι ο θεματοφύλακας των διαδικασιών. Είναι σημαντικό να έχουμε διαδικασίες όμοιες σε όλη την Ευρώπη και ε, χρειάζεται μια εξελικτική προσέγγιση προς την ευρωπαϊκή ε, αδειοδότηση των οχημάτων. Ε, θα υπάρχει συνεργασία με τον ΕΟΣ και είναι σημαντικό να πούμε ότι ο ΕΤΟΝ ορίζει τον τομέα χρήσης ε, που θα λειτουργούν τα τρένα και ο τομέας χρήσης θα καλύπτεται από την αδειοδότηση των οχημάτων απόλυτα. Όταν οριστεί ο τομέας της λειτουργίας τότε θα υπάρξει αδειοδότηση για το συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης, η τωρινή πρόταση της Κομισιόν είναι συμβατή με όλα τα παραπάνω και τις προτεραιότητες του τομέα και, του τομέα και νομίζουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν ως έχει. Και για να τελειώσω... Τρεις βασικές ιδέες. Ο κλάδος των σιδηροδρόμων χρειάζεται εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αδειοδότηση των οχημάτων. Πρέπει όλα να ε, είναι ε, συμβατά, ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία και ο τεχνικός πυλώνας του, της, τέταρτης, δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους δεν θα πρέπει να επιβραδυνθεί ή δυνατόν και ε, ε, δεν θα πρέπει δηλαδή να επιβραδυνθεί από άλλα κομμάτια της ε, δέσμης μέτρων. Αν υπάρχουν άλλα τμήματα θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Θα πρέπει οι μηχανικοί μας να δουλέψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα και να μην δαπανούν ώρες επί ωρών για την αδειοδότηση των οχημάτων. Οι μηχανικοί μας, οι μηχανολόγοι θα πρέπει να δουλέψουν για ένα ευρωπαϊκό μέλλον και να αφιερωθούν στον δικό τους τον κλάδο, στα μηχανολογικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε. Διότι να, ευχαριστ... να καλωσορίσω ταυτόχρονα στην Επιτροπή μου 40 φοιτητέ από το Collège de France της Μασαλίας μετά από πρόσκληση του των Συγγνώμη που σας ε, έχουμε να στέκεστε. Το πρόβλημα με το Κοινοβούλιο είναι ακριβώς η πρόσβαση στις συναντήσεις ε, των επιτροπών όπου θα μπορείτε να κάτσετε και να παρακολουθήσετε. Αυτό είναι ατυχές αλλά χρειάζεται να κρατήσουμε θέσεις για τα μέλη εδώ οπότε συνήθως τα υπόλοι, οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από τα λόμπι. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη που είσαστε υποχρεωμένοι να στέκεστε όρθιοι. Πάντως είσαστε ευπρόσδεκτοι. και υγιές φορές πραγματικά απελπίζομαι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κοινό που έρχεται στις συναντήσεις μας και τους βάζουμε να στέκονται όρθιοι ακουμπισμένοι στους τοίχους το πίσω μέρος της αίθουσας. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε. Ίσως θα έπρεπε να το δουν οι υπεύθυνοι του Κοινοβουλίου δεν έχουμε θεωρία επισκεπτών, θεωρία δημοσίου. Θέλετε να δείτε να κάτσετε, μπράβο Μάικλ, δίκιο έχεις. Ελάτε να καθίσετε εδώ πέρα. Εκεί που έχετε τις πράσινες πινακίδες. Πραγματικά είναι γελίο. Αλλά άμα θέλετε ελάτε. Ξέρετε ότι θα κάτσετε όλο το απόγευμα. Και όπου βλέπετε πράσινο καρτελάκι καθίστε. Και αν σας πει κανείς τίποτα να τους πείτε ο πρόεδρος μου το είπε. Και μπροστά μπροστά στην πρώτη σειρά μα θέλετε ελάτε. Υπάρχουν στην πρώτη σειρά εννέα άδειες θέσει γιατί βαριούνται να κάτσουν στην πρώτη σειρά γιατί πιάνει το σβέρκος τους.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 Here you are, young ladies. Here you are. Down here. Yeah. Yeah, yeah. There we go. Ωραία. Λύσαμε το πρόβλημα Πραγματικά μου τη σπάει το μερά αυτό το πράγμα. Διότι έρχονται όλοι τα λόμπι και λένε ότι εκπροσωπούν τους πολίτες, ε, ότι εκπροσωπούν τους πολίτες ε, της Ευρώπης και έρχεται ένας πολίτης και στέγεται όρθιος ο Κακομύρης. Λοιπόν, από την προοπτική των ε, επιχειρήσεων, ο κ. Σάιντχόβεν, συγγνώμη που καθυστέρησα, από την Netherlands for Spolang και τους Ολλανδικούς Συνδεδρόμους ο κύριος Βαν Άιτχόβεν. Φορέστε τα ακουστικά σας εσείς στα γαλάκια, στα, στο τρία είναι. Κύριε Άιτχόβεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ΕΝΕΣ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να μιλήσω στην Επιτροπή Μεταφορών για τόσο σημαντικά θέματα της Ένωσης. Μου ζητήσετε, Πρόεδρε, να σας ε, δώσει η εταιρεία μου, η τους στόχους, την άποψή της για τους στόχους που έχουμε επιτάπτει. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά να σας πω εντάχει τι πετύχαμε για τις συνδρομικές μεταφορές στην Ολλανδία. Μετά το πρώτο συνδρομικό πακέτο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, η Ολλανδία θέτησε τους κανόνες γρήγορα. Κάτι που εφαρμοζόταν και για το επόμενα πακέτα. Και αυτό έδωσε αποτελέσματα. Οι διαχειριστές των υποδομών και οι μεταφορείς διαχωρίστηκαν, αλλά προς το συμφέρον των επιβατών έγινε, ξεκίνησε μια εντατική συνεργασία μεταξύ των δύο. Χάρη στην ε, απελευθέρωση που έγινε, η μεταφορά, οι εμπορευματικές μεταφορές είναι τελείως ελεύθερα, ενώ οι επιβατικές προχωρούν προς την ε, απελευθέρωση. Το ένα είναι ο μεγαλύτερος μεταφορέας στην Ολλανδία, με κάπου 140 εκατομμύρια τρένο, τρένο χιλιόμετρα καλύπτονται κάθε χρόνο. Ενώ άλλα 25 εκατομμύρια καλύπτονται από όλους φορείς σε 30 διαδρομές. Η ΕΝΕΣ έχει παίξει έναν όλο και μεγαλύτερο εμπορικό ρόλο. Οι εκχωρήσεις που μας έδωσαν η, μας έδωσε η κυβέρνηση εγκαταλείφθηκαν προς, ε, προς όφελος άλλων μορφών συμπληρωματικών μεταφορών. Είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια αύξηση 10% στον αριθμό της, μεταφορά, της μεταφοράς επιβατών. Αποτέλεσμα μετά μιας δεκαετίας υλοποίηση του συνδρομικού πακέτου στη χώρα μου. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι το τέταρτο πακέτο δεν πρέπει να το βλέπουμε χωριστά από τα προηγούμενα. Ο κύριος στόχος του είναι να ο κίνδυνος να, πάθει, να, να υποστεί ο Ολλανδικός Ιδεόδρομος μια υποχώρηση. Αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά χρειάζεται, χρειάζονται νέες ε, βελτιώσεις. Η απάντησή μου είναι και ναι και όχι. Τεχνικά η Επιτροπή κάνει μια σειρά προτάσεων και η ΕΝΕΣ θεωρεί ότι αυτό έχει πολλά θετικά στοιχεία. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη, να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικά τα πράγματα, να δουλέψουμε για πιο σύγχρονου ιδιοδρόμου και να κάνουμε αυτό το modal shift που απαιτεί η Ευρώπη. Αυτή είναι η άποψή μας για τον κανονισμό PSO, αλλά φοβόμαστε ότι το τέταρτο πακέτο πραγματικά δεν προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση αυτή. αυτό θέλω, γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω τις θέσεις του NS. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω καταρχάς για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Συνδρομική Υπηρεσία, το ERA. Η κατάσταση έτσι όπως περιγράφεται, μας καλύπτει. Οι διαδικασίες πιστοποίησης του τοχείου υλικού σήμερα είναι μεγά, μακροχρόνιες και δαπανηρές. Προφανώς οι εθνικές ε, και αρχές ασφάλειας θα πρέπει να, παίξουν, να συνεχίζουν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουν πώς λειτουργούν οι υποδομές και το επίπεδο ασφάλειας. Οι γνώσεις τους είναι αναγκαίες, κρίσιμες για την οσιοδρομική ασφάλεια και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί. Ωστόσο, ο ρόλος που προβλέπεται για την αίρα ως one-stop shop για όλους τους μεταφορείς και συντονιστές θα διευκολύνει τις αιτήσει και θα επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης. Ε, εάν οι αλλαγές αυτές υλοποιηθούν ουσιαστικά θα είναι για την κατάποψή μας ένα βήμα μπρο. Επίσης, θέλουμε πολύ θετικές τις προτάσεις της Επιτροπής για την διαλειτουργικότητα. Η ίδια η Ολλανδία είχε περιγράψει ένα rail map για το ERTMS με βάση την εμπειρία που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Η ΕΝΕΣ μετέχει στις εξελίξεις και συζητήσεις και βλέπει τους περιορισμούς, τους υφιστάμενους περιορισμούς στην αγορά, όπως την απουσία προ, προτύπων για ανοιχτά ETCS και για την μονοπωλιακή θέση κάποιων ε, προμηθευτών. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΑΕΡΑ για τα, την άδεια ERTMS. Το πλαίσιο αυτό θα, στο πλαίσιο αυτό το ΕΡΑ θα πρέπει να δημιουργεί τους βέλτιστους ε, δυνατότητες, βέλτιστες δυνατότητες για να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες προφανώς. Στις, ε, η, στην Ολλανδία η χωρητικότητα του δικτύου είναι βασικό θέμα, θέμα και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη η νέα νομοθεσία. Στη νέα πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ERA, το άρθρο 24 ορίζει τον ρόλο της ERA σαν μια συστημική αρχή για το ERTMS. Ο ρόλος αυτός, ο κεντρικός ρόλος για την υλοποίηση του ERTMS γίνεται σημαντικότερος ε, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι ΕΝΕΣ θεωρούν ότι αυτή η συστημική ο συστημικός ρόλος του ΕΡΑ, e είναι, του ΕΡΑ e είναι που θα επιτρέψει να προχωρήσουμε. Τώρα, για τον κανονισμό PSO υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και για τους, ε, μεταφορικούς τους ε, φορολογούμενους και για τους, και ταξιδιώτες. Γιατί το, το σύστημα αυτή τη στιγμή εμποδίζει την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Γιατί αυτό. Λόγω των περιορισμών στα PSO, οι περιορισμοί έχουν αρνητικές επιπτώσεις και δεν συμβάλλουν όπως προϋποθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν πλέον να οργανώσουν μόνο τους την κινητικότητα. Οι περιορισμοί στον όγκο για τις ε, επιβατικές μεταφορές που προκύπτουν από μία άδεια, χωρίς να, λάβει, να λάβουμε υπόψη την ειδική κατάσταση της κάθε χώρας, θα οδηγεί στην Ολλανδία σε τρίχα, σε μία διέρισε τρία τμήματα του δικτύου, κάτι που θα είναι κακό για τους ε, επιβάτες. Το εφιστάμενο σύστημα που είναι και ενοποιημένο και βελτιστοποιημένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύστημα λιγότερο θετικό και που θα πετύχει μεγαλύτερο συντονισμό, μεγαλύτερη ρυθμισή και θα θέσει σε κίνδυνο όλα τα πλονεκτήματα της απελευθέρωσης. Είναι μια περιττή εμπλοκή του κράτους που μετατρέπεται χωρίς να το θέλουμε σε επιχειρηματία. Λόγω αυτής της ε, μείωσης της αποτελεσματικότητας αναμεταφορέ οι επιβάτες θα χρειαστεί να αλλάζουν συχνά τρένα, κάτι που δημιουργεί προβλήματα και η ενώ η εγκατάλειψη κάποιων γραμμών θα αποδυναμώσει το κοινό. Η υφιστάμενη υποδομή και οι υφιστάμενες υπηρεσίες είναι απόλυτα εναρμονιμένες. Αυτό επέτρεψε στην Ολλανδία να έχει σημαντική αύξηση της χρήσης των υποδομών. Ο κατακαιρματισμός του υφιστάμενου δικτύου θα οδηγήσει σε υποχώρηση και της ποιότητας και των υπηρεσιών προς τον ταξιδιώτη. Θα ήταν επίσης κακό και για τον ε, φορολογούμενο, διότι ε, ο κατακαιρματισμός του δικτύου μεταξύ πολλών θα απαιτήσει μεγαλύτερες επενδύσεις, κάτι που δεν θέλει η κυβέρνηση. Το έχει πει ο υπουργό ήδη. Η υποδομή που σε κάποια κομμάτια του εδάφους είναι ανεπαρκής δεν θα χρησιμοποιείται επαρκώς, ενώ τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται περισσότερο δεν θα έχουν χώρο για επιπλέον τρένα. Με άλλα λόγια, η πρόταση της Επιτροπής στο θέμα αυτό έχει μόνο ανατρεπτικά αποτελέσματα. Μόνο επιπλέον επενδύσεις σε υποδομές που θα επέτρεπαν, ενώ οι επενδύσεις μάλλον στις υποδομές δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα, οικονομικά, τα, τα μέτρα. Η μάχη κατά των ανισοτήτων και των κενών αυτών απαιτεί περαιτέρω επένδυση από το κράτος και άρα αύξηση του κόστους για τον φορολογούμενο. Να τελειώσω. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την απελευθέρωση ήδη από το πρώτο πακέτο. Τα μέτρα, με τα μέτρα για τον αέρα και την διαλειτουργικότητα θα ενισχυθεί περαιτέρω ο τομέας εφόσον οι νέες ευθύνες αναλυθούν και ελέγχονται, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι ευθύνες των εθνικών αρχών ασφάλειας. Με άλλα λόγια, οι ΕΝΕΣ θεωρεί θετικές τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, ιδίως τεχνικά. Η πρόταση η απελευθε, ότι η απελευθέρωση του συνδρομικού κλάδου στην τομέα δεν έχει ε, αποτελέσματα είναι λάθος, κατά την άποψή μας τουλάχιστον και δεν ισχύει για, την για τη βορειοδυτική Ευρώπη τουλάχιστον. Οι προτάσεις για το PSO, ωστόσο, είναι κακές για ένα δίκτυο όπως αυτό της χώρας μου. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με μεγαλύτερη απορρίθμιση των σιδηροδρόμων, αλλά είμαστε αντίθετοι με τον κατακαιρματισμό που θα είναι και αυθαίρετος. Αυτό θα ήταν κακό για τους επιβάτες και για τον φορολογούμενο στην Ολλανδία. Η ενιαία προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή ήταν κακό εργαλείο για την επίτευξη ενός ε, αξιέπαινου στόχου. Η ΕΝΕΣ υποστηρίζει την μελέτη του δικού μας ε, Υπουργείου να έχει κάθε χώρα δικό της πλαίσιο ε, για τι ιδεοδοτικέ μεταφορέ και να έχει δικό τη στόχο για να, το, να πετύχει του στόχου που θέλει η Επιτροπή. Αυτή η ελευθερία επέτρεψε ακριβώ την ανάπτυξη του ιδεοδομικού δικτύου στην Ολλανδία και την αύξηση και των επιβατών και του κύκλου εργασιών. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή θα μας εκφράσει την πανεπιστημιακή προοπτική, την πανεπιστημιακή πλευρά. Πρόκειται για τον Ερνέστο Γκαρθία Βαντίλο, καθηγητή στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της χώρας των Βάσκων από την Ισπανία. Έχετε το λόγο. Για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την άποψη ενός πανεπιστημιακού. Η παρουσίασή μου δεχίστε παρακαλώ, ο Πρόεδρος. Η παρουσίαση μου εστιάζεται στην αναθεώρηση των προτάσεων διαλειτουργικότητας. Καταρχάς θα θέλω να πω κάποια πράγματα για την ίδια την οδηγία, για τον επαγγελματικό μας κλάδο, καθώς επίσης και τους διαχειριστές υποδομής Στη συνέχεια θα αναφερθώ στα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στην οδηγία. Τρίτον, θα αναφερθώ στο ζήτημα της διαλειτουργικότητας, καθώς επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. Τέταρτον, θα αναφερθώ στα εκρεμή ζητήματα που υφίστανται στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και θα αναφερθώ επίσης και στην επίδραση που έχουν όσον αφορά τις πανεπιστημιακές μελέτες που γίνονται. Και τέλος θα προσπαθήσω να δείξω πώς οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές λειτουργικότητας πρέπει να σωματωθούν με τεχνικά πρότυπα. Και θα καταλήξω έπειτα σε κάποια συμπεράσματα. Για έναν εξωτερικό ανεξάρτητο παρατηρητή φαίνεται σαφές ότι η οδηγία αυτή θα ευνοήσει τους κατασκευαστές, όπως το ακούσαμε πριν από λίγο, καθώς επίσης φαίνεται ότι προστατεύει και τους διαχειριστές υποδομών, τουλάχιστον στο άρθρο 11 σημείο 1, μπορεί να βάσει κανείς ότι όποτε ένα κράτος μέλος συντοπεί ότι ένα συστατικό στοιχείο εξάρτημα της υποδομής δεν καλύπτει τη δήλωση συμμόρφωσης, θα μπορεί να αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσει το πεδίο χρήσης του και εφαρμογής του, να απαγορεύσει τη χρήση του, να το αποσύρει από την αγορά. Να πω κάποια πράγματα όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα τώρα. Στην πρόταση συγκεκριμένα στο άρθρο 29 σημείο 1 λέγεται ότι το προσωπικό το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, καθώς επίσης και την επαλήθευση θα πρέπει να έχει μια πολύ καλή τεχνική και επαγγελματική προετοιμασία προκειμένου να αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί Πρέπει να σας πω ότι ο κλάδος αυτός των σιδηροδρόμων από μηχανικής πλευράς είναι τεράστιος, πάρα πολύ ευρύς. Και δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα για πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι μηχανικοί σε ζητήματα σιδηροδρόμων. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Για παράδειγμα, η δυναμική των σιδηροδρόμο όσον αφορά την ταχύτητα μπορεί να αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχουν μάλιστα και πολλά πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν σπουδές πολύ ψηλού επίπεδου προκειμένου να μπορεί κανείς να εξειδικευτεί και να ανταποκριθεί στι απαιτήσει του σιδηροδρομικού τομέα. Περνώ τώρα στο επόμενο σημείο της παρουσίασής μου, στο οποίο θα αναφερθώ στην διαλειτουργικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι ακριβώς γίνεται με τα TSI, με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Δεν απαιτώ από εσά να διαβάσετε όλα αυτά τα οποία αναφέρω στη διαφάνειά μου, να αναφέρω απλώς ότι υπάρχουν 17 τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, 5 εκ των οποίων είναι εγκάρσιες, οι υπόλοιπε 5 αφορούν τα τρένα υψηλή ταχύτητα και οι υπόλοιπε 7 αφορούν του συμβατικού σιδηροδρόμου. Τρει λοιπόν από τι τεχνικέ προεγγραφέ λειτουργικότητα τι έχω σημειώσει με ένα βέλο στην παρουσίασή μου και θα ήθελα να σα πω πω για τι περισσότερε από αυτέ υπάρχουν ακόμα κάποια εκκρεμή ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Και νομίζω ότι εδώ πέρα μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο οι καθηγητέ πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα υποσυστήματα υποδομή, υπάρχουν τέσσερα εκκρεμή ζητήματα. Πρώτον, απαιτήσει για τον έλεγχο τη ισοδύναμη κονικότητα απαιτήσει όσον αφορά τα προβλήματα της καμψίας της τροχιάς και αυτό το ζήτημα παραμένει εκρεμές. Έχουμε επίσης προβλήματα δονήσεων καθώς επίσης και θορύβου και πώς μπορούν να μειωθούν τα φαινόμενα αυτά από πλευρά υποδομής και τέλος έχουμε και κάποιες απαιτήσει για την μείωση των επιπτώσεων των πλευρικών ανέμων. Όσον αφορά το τροχαίο υλικό τώρα, και εδώ πέρα έχουμε πάλι ένα ανοιχτό, ζήτημα όσον αφορά την παρακολούθηση του λιποκιβωτίου άξονα. Προβλήματα επίσης έχουμε με τους άξονες μεταβλητού εύρους. Και όσον αφορά τις μηχανές και όσον αφορά το τροχείο υλικό για τους επιβάτες, υπάρχει ένα γενικότερο εκκρεμές ζήτημα που έχει να κάνει με το όλο σιδηροδρομικό δίκτυο και ορισμένα τα οποία μπορούν να κατηγοροποιηθούν με βάση την τεχνική συμμόρφωση που υπάρχει ανάμεσα στο δίκτυο και το όχημα και κάποια άλλα κρεμή ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τεχνική συμμόρφωση μεταξύ οχήματος και δικτύου. Θα σας δώσω τώρα δύο παραδείγματα. Δύο πραγματικά παραδείγματα. Ελπίζω να μην ξανασυμβούν ποτέ, να μεταξύ να δούμε μπροστά μα, αλλά δείτε για παράδειγμα τη διαφάνεια αυτή. Βλέπετε εδώ πέρα ποιε είναι οι επιπτώσει τη χρήση μια παλιά διζελομηχανή. Βλέπετε εδώ πέρα ποιε ήταν οι επιπτώσει στην σιδηροδρομική τροχιά μετά το πέρασμα τη μηχανή αυτή. Α αποφύγουμε τέτοια παραδείγματα στο μέλλον προφανώ. Α δούμε ένα ακόμα παράδειγμα. Επιπτώσει τη χρήση ακατάλληλου σιδηροδρομικού υλικού, το οποίο προκάλεσε φθορά κεφαλής του άξονα. Διάβρωση την οποία βλέπετε στη διαφάνεια αυτή. Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αποφευχθεί. Και σας πω τώρα ότι υπάρχει μία πρωτοβουλία η οποία ονομάζεται Shift to Rail στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 ο οποίο αρχίσει να ισχύει μετά το 7ο πρόγραμμα έρευνα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι θα πρέπει προφανώ να προωθήσουμε τον ορίζοντα 2020, καθώ επίση και τα επιμέρου προγραμματά του, όπω το SHIFT του RAIL. Βλέπετε εδώ πέρα πέντε ερευνητικέ προτεραιότητε, οι οποίε έχουμε εντοπίσει επαρκής τεχνολογίας όσον αφορά τα τρένα υψηλής χωρητικότητας, προηγμένα συστήματα διαχείρισης ε, των δικτύων και των συστημάτων ελέγχου, καλύτερες τεχνολογίες όσον αφορά τα, ε, τους βιώσιμους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, καθώς επίσης και λύσεις όσον αφορά την άρρηκτη ε, διασύνδεση των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας και τα εθνικά πρότυπα. Επί του παρόντος έχουμε τα εθνικά πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας, καταλαβαίνετε ότι οι εθνικοί οργανισμοί που καταρτήσουν τα εθνικά πρότυπα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων κάποια στιγμή θα πρέπει να συγχωνευτούν. Επίσης έχουμε πανεπιστήμια σε κάθε κράτος μέλος που θα μπορούσαν ανεξαρτήτως να βοηθήσουν να επιτευχθεί η ενσωμάτωση αυτή και η ομογενοποίηση αυτή την οποία θέλουμε να πετύχουμε και να περάσω τώρα στα συμπεράσματα της παρουσίασής μου. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το σχέδιο οδηγίας ευνοεί τους, κατασκευα... κατασκευαστές και επίσης εξετάζει το πώς μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τους διαχειριστές υποδομών. Δεύτερο συμπέρασμα, ένα σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ήδη δραστηριοποιούνται πάρα πολύ σε συγκεκριμένη εκπαίδευση όσον αφορά την τεχνολογία σιδηροδρόμων και είναι σε θέση να παρέχουν, να καταρτήσουν καταρτισμένο προσωπικό. Έπειτα έχουμε την πρωτοβουλία Shift to Rail στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Ορίζοντας 2020. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεματικό πρόγραμμα, μια θεματική πρωτοβουλία που μπορεί να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα που έχουμε στα πλαίσια των TSI. Αναφέρθηκα σε ορισμένα, αλλά υπάρχουν και πολλά περισσότερα. Και νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή χρειάζεται μια ενεργή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από, τις επιτροπές, από την Επιτροπή Μεταφορών και Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έπειτα θα ήθελα να προτείνω το να κινητοποιηθούν περισσότερο τα πανεπιστήμια στα κράτη-μέλη, γιατί είναι σε θέση ως ανεξάρτητοι φορείς να βοηθήσουν την ενσωμάτωση των TSIS και των εθνικών προτύπων. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκαρθιά Βαντήλο. Επόμενος ομιλήτης ο κύριος Μίκο Πέρις, ο οποίος ε, είναι project manager των Βαλτικών Σιδηροδρόμων στο Εστονικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών. Ο κύριος Πέρις έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, όπω αναφέρθηκε, λέγομαι Μίκο Πέρι και εργάζομαι για το Εσθονικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών και είμαι ο Εσθονό Project Manager ενό σημαντικού περιφερειακά σιδηροδρομικού έργου στο σιδηροδρόμου τους Βαλτικού. Σήμερα θέλω να παρουσιάσω την άποψη των εμπειρογνωμών σχετικά με τον κανονισμό, σχετικά με τι νέε αρμοδιότητε του ΕΟΣ, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ΕΟΣ θα τον λέμε. Ε, προέρχομαι από την Εστονία, αλλά ε, θα μιλήσω με ευρύτερο, σε ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο για τις βαλτικές χώρες γενικά. Είναι γνωστό ότι τα σιδηροδρομικά συστήματα των βαλτικών κρατών διαφέρουν λίγο από την, εκείνα της υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, Για ιστορικούς λόγους το δίκτυο το σιδηροδρομικό μας τώρα δεν είναι συνδεδεμένο απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Γι' αυτό το βαλτικό δίκτυο πολλές φορές αναφέρεται ως απομονωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο και αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε πολύ όταν συζητάμε για τις νέε αρμοδιότητες του ΕΟΣ. Παράλληλα όμως υπογραμμίζω ότι τίποτα στην ομιλία αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη συμφόρηση. Αντίθετα, η νέα γραμμή των βαλτικών σιδηροδρόμων που θα κατασκευαστεί θα ε, πληρώσει το κεμνό στο ευρωπαϊκό δίκτυο διευρωπαϊκών ε, δικτύων μεταφορών και Τώρα όλες οι βαλτικές χώρες με την Πολωνία και τη Φιλανδία κάνουν κοινέ προσπάθειες για να, γίνει το, να γίνουν οι βαλτικοί σιδηρόδρομοι ολοκληρωμένοι μέχρι το τέλος του 2023. Κυρίε και κύριοι, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η Κομισιόν υπέβαλε καλό πακέτο. Η τέταρτη δέσμη ε, είναι πάρα πολύ σημαντική δέσμη γιατί οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ιδηροδρομικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κερδίσει πολλά από την έκβαση αυτού της δέσμης μέτρων. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς κατά των βασικών αξώνων του της δέσμης που είναι άνοιγμα τη αγορά σιδηροδρόμων, εναρμόνιση των κανόνων διαλειτουργικότητα και ασφάλεια και τέλο, αλλά πολύ σημαντικό, μείωση τη γραφειοκρατία στη διαδικασία επιστοποίηση. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά σίγουρα είναι ευπρόσδεκτα και είναι αναγκαίοι στόχοι. Πιστεύουμε δε ότι οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί θα συμβάλλουν πραγματικά στη λειτουργία μιας ευρωπαϊκής κοινής αγοράς γενικότερα και στην ενιαία, στον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο ειδικότερα. Τώρα θα μιλήσω για τι λεπτομέρειε του προτινόμενου σχεδίου κανονισμού σχετικά με τι αρμοδιότητε του ΕΟΣ. Θα κάνω τρει βασικέ παρατηρήσει και μετά θα ε, αναδείξω ε, κάποιε πιθανέ πιθανές ε, βελτιώσεις. Καταρχήν, θέλουμε καλύτερο καταμερισμό εργασίας μεταξύ των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας και του ΕΟΣ. Τώρα, το, οι δέσμοι μέτρων ε, παρουσιάζει έναν κατακαιρματισμένο μάλλον κατάλογο καθηκόντων για τους ε, αρμόδιους ε, φορείς. Έτσι είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και να καταλάβουμε ποιες υποχρεώσεις και καθήκοντα έχουμε για τη μέγιστη ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Πώς θα συμβάλλουμε και εμείς αυτό. Χαιρετίζουμε τις επιμερισμένες αρμοδιότητες μεταξύ του ΕΟΣ και των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας και πιστεύουμε ότι η νομοθεσία θα πρέπει ε, σαφέστατα και να εξπρέσεις βέρμπης να προβάλλει εξαντλητικό κατάλογο των καθηκόντων αυτών των δύο φορέων. Ε, προφανώς ένας στόχος πρέπει να είναι να αποφεύγουμε επικαλύψεις εργασιών και να διασφαλίσουμε ε, καλά ισορροπημένο καταμερισμό εργασίας. Ως μέρος του καταμερισμού αυτού εργασίας η συγκεκριμένη περίπτωση των μεμονωμένων δικτύων μπορεί να ληφθεί υπόψη. Για παράδειγμα, ο καταμερισμό εργασία στο τομέα τη πιστοποίηση μπορεί να στηρίζεται στο αν οι ε, σιδηρόδρομοι θα τα τρένα θα χρησιμοποιηθούν στο ευρωπαϊκό δίκτυο με το συγκεκριμένο του εύρος, ε, δηλαδή 14-35 ε, έχει λιωστά δίκτυο ή το άλλο. μια λύση είναι ο ΕΟΣ να παίξει το ρόλο της μόνο υπηρεσίας συντονίζοντας τις αρμόδιες αρχές, εθνικές αρχές ασφάλειας. Αλλά αν το όχημα χρησιμοποιείται μόνο σε ένα, θα χρησιμοποιείται μόνο σε ένα κράτος μέλος, ο ετών μπορεί να διαλέξει μεταξύ του ΕΟΣ και των αρμόδιων, της αρμόδιας εθνικής αρχής ασφάλειας. Η αδειοδότηση τροχαίου υλικού που προτίθεται να χρησιμοποιηθεί για, ε, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο Εκεί η πιστοποίηση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική ε, στα χέρια των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας. Ως γενική, ε, γενικός κανόνας όμως ε, είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι ο ΕΟΣ θα αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο και ευθύνη στον τομέα της πιστοποίησης και εμείς θέλουμε να επιτευχθεί ο στόχος της Κομισιόν για την εναρμόνιση και την επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης σε όλη την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, μετά τον καταμερισμό εργασία πρέπει να είναι σαφής, θα πρέπει να έχει ο ΕΟΣ ε, σαφείς εξουσίες ε, να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο επί των αρχών ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ΕΟΣ θα πρέπει να έχει σαφή νομική βάση για να παρεμβαίνει, είτε φαίνεται ότι ε, δεν κάνουν καλά τα καθήκοντά τους οι εθνικές αρχές ή τίποτε άλλο. Αν μπορεί να υπάρχουν δηλαδή ε, καθυστερήσεις άσκοπες και τότε η προσφυγή, η καταγγελία θα γίνει από τη συνδρομική επιχείρηση κλπ. Ειδικότερα η αρχή του ΕΟΣΕ επί των εθνικών κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας θα πρέπει να προστατεύεται και όπως προβλέπεται ήδη στο σχέδιο κανονισμού. Σίγουρα χαιρετίζουμε τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ του ΕΟΣ και των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας. Τρίτον, προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι αρμοδιότητες του ΕΟΣ να αυξηθούν με βάση τη σταδιακή προσέγγιση και να γίνει ένα phasing in σταδιακή δηλαδή ε, διεύρυνση. Το τελευταίο θα πρέπει να γίνει με σαφή ορόσημα και λεπτομερείς διατάξεις μεταβατικές που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία. Αυτό γιατί στην αρχή ο ΕΟΣ είναι πιθανόν να στηρίζεται στο έργο των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας στην πρώτη φάση και λόγω των τεχνικών ε, προτύπων διαλειτουργικότητας που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εμεί πιστεύουμε ότι καλό θα είναι να τεθεί μια βέλτιστη μεταβατική περίοδο μέχρι ότου τεθούν σε ισχύ αυξημένε αρμοδιότητες του ΕΟΣ. Επίσης πρέπει να πω ότι τώρα οι Εθνικές Αρχές ασφαλεία στις χώρες της Βαλτική έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στο ρόλο τους και σε ό,τι αφορά το χρόνο και το χρήμα. Η αποτελεσματικότητα πρέπει να διατηρηθεί και να γίνει το modus operandi του ΕΟΣ όταν αναλάβει το νέο ρόλο του ο τελευταίο. Ε, θα προτείναμε για την αποτελεσματικότητα να υπάρχει ένα συνεκτικό σύστημα ενημέρωσης ε, τεχνολογίας πληροφοριών το οποίο θα έχει στόχο να εξυπηρετεί τις διαδικασίες πιστοποίησης και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνοψίσω την άποψη των βαλτικών χωρών για τον κανονισμό του ΕΟΣ. Εμείς βλέπουμε την αξία των αυξημένων αρμοδιοτήτων του ΕΟΣ, όμως ε, επειδή υπάρχουν πολλές ανισότητες ε, και διαφορές στη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο, θέλουμε σταδιακή προσέγγιση στην αύξηση των ε, αρμοδιοτήτων του ΕΟΣ. Επίσης θέλουμε να είναι σαφής η διατύπωση που σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ του ΕΟΣ και των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας. Ως μέρος αυτού του καταμερισμού εργασίας ζητούμε αναλογική η κατανομή αρμοδιοτήτων που θα τύχει επεξεργασία σε επίπεδο κρατών μελών ε, που έχουν μεμονωμένα δίκτυα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ε, αποτελεσματικές διαδικασίες πιστοποίησης από το νεό στο μέλλον. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε και παραμένουμε στην διάθεση της Επιτροπής Μεταφορών για μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής από την οπτική των ε, υπεύθυνων διαχείρισης, ο κύριος Διενόδη, για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να τηρήσω το... Να σας πω γιατί θα μιλήσω. Το Steve Davis Gleave ανέλαβε την διεξαγωγή των μελετών υποστήριξης του τέταρτου πακέτου Μία από τι μελέτε είχε να κάνει με το μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, του Ευρωπαϊκού Συνδρομικού Οργανισμού, τη τεχνική διάσταση του Ευρωπαϊκού και αυτό θα είναι ε, το βασικό σημείο τη παρουσίασή μου σήμερα. Όταν κάναμε το έργο που είχαμε αναλάβει, βασική παράμετρος ήταν να τηρήσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μελέτη αντικτύπου και να τηρήσουμε τις απαιτήσει της Επιτροπής για όλες τις μελέτες αντικτύπου. Γι' αυτό αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η λεπτομεριακή ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων, να μιλήσουμε δηλαδή με όλους με πολλούς από εσά που είστε εδώ σήμερα και με άλλους για να ακούσουμε την άποψή σα για τον καλύτερο μελλοντικό ρόλο του οργανισμού και να αναπτύξουμε την ανάλυση μέσω του εντοπισμού των βασικών προβλημάτων προτείνοντα ε, συγκεκριμένε πολιτικέ που πρέπει να ακολουθούν. ακούσαμε ήδη πολλά από τα προβλήματα ειδικά για τις διαστάσεις που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα. Είδαμε ωστόσο και εδώ το πρώτο, η πρώτη κουκίδα είναι οι τεχνικές, οι δυσκολίες ε, και τα διοικητικά εμπόδια. Πρόκειται για μια μακρά πρόταση που καλύπτεται ωστόσο, που καλύπτει τέσσερις τομείς. Πρώτον, ανεπαρκή λειτουργία των εθνικών θεσμών. Διακριτική αντιμετώπιση των εισερχόμενων από εθνικού φορεί. Διαφορετική ερμηνεία της Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία και η κληρονομιά των εθνικών σιδηροδρομικών συστημάτων. Πρώτον, η λειτουργία των εθνικών δομών οι πληροφορίες που πήραμε από πολλούς εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων την ίδια, την, τον ίδιο τον Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Μηχανισμό, μας έδωσε να διαπιστώσουμε μια σειρά διαστάσεων που πρέπει να δούμε λεπτομεριακά σε σχέση με τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τις πρακτικές τους. Πρώτη είναι οι πόροι που, έχει στη διάθεση του, που έχουν στη διάθεσή του οι εθνικέ αρχέ ασφάλεια σήμερα. Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση στο προσωπικό που ασχολείται με θέματα διαλειτουργικότητα από ένα άτομο σε 162. Επίση, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στου πόρου, στους οικονομικού πόρου που διατίθενται στι ε, υπηρεσίες αυτές. Το κόστο του πιστοποιητικού ασφάλεια, ποικίλει σημαντικά. Σε κάποια κράτη δεν υπάρχει κόστος. Σε άλλα το κόστος μπορεί να φτάσει να ξεπεράσει τα 70 χιλιάρικα. Προφανώς στην Ευρώπη το 15 το μέσος όρος είναι υψηλότερος, αλλά υπάρχει μια εικόνα ότι και στις νέες χώρες, τις 12 αυξάνεται. Επίσης, η, η αδειοδότηση των οχημάτων. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στο κόστος της ε, Έγκριση των οχημάτων. 1,6 εκατομμύρια ένα όχημα λέει η ΕΡΑ, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια. Πέραν του κόστους δε υπάρχει και ο χρόνος που έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Βλέπετε εδώ το παράδειγμα 10 ε, έως και 90 εργάσιμων ημερών για ε, εμπορευματικά οχήματα. Οπότε όταν βλέπουμε ολόκληρα, ολόκληρες σειρμούς θα δείτε ότι μιλάμε για τεράστια... Για παράδειγμα, για ένα τρένο μας αναφέρθηκε περίπτωση όπου ένα τρένο καθυστέρησε 7 χρόνια η αδειοδότησή του. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποιο που θέλει να κάνει επενδύσει δεν μπορεί να προγραμματίσει πότε θα ξεκινήσει η υπηρεσία. Προφανώ οι εμπλεκόμενοι που συζητήσαμε θεωρούν πολύ ψηλό το κόστος και πολύ μεγάλο το χρόνο. Συχνά η κατάσταση επιδεινώνεται, είναι χειρότερη για τους νεοεισερχόμενους. Μιλήσαμε με κάποιους νεοεισερχόμενους, όχι όλους, Κάποιοι μα είπαν ότι θεωρούν πως πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν με διακριτικό τρόπο από τι εθνικέ αρχέ στη διαδικασία πιστοποίηση και έγκριση. Και εγώ μιλώ για νοησερχόμενους, όχι μόνο για νοησερχόμενους που μπαίνουν στην εθνική αγορά, αλλά και για νεοεισερχόμενους που μπορεί να είναι οι παλιοί, οι εγκατεστημένοι, εγκατεστημένοι άλλου κράτου μέλους που μπαίνουν σε νέα αγορά. Αυτό δημιουργεί σοβαρά εμπόδια εισόδου που δυσχερά ενώνει την δημιουργία αυτού του ευρωπαϊκού ενιαίου χώρου μεταφορών. Επίσης, βλέπουμε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας διαφοροποιείται σημαντικά. 62% των εμπλεκόμενων με τους οποίους μιλήσαμε θεωρούν ότι αυτό είναι πρόβλημα. Το ποσοστό που βλέπετε στην οθόνη από αριστερά προς δεξιά αναφέρει πρώτον τα κράτη-μέλη που, που δεν ανέφεραν καθόλου με μηδέν και τα κράτη-μέλη σε όλο και μεγαλύτερη αύξηση που αναφέρουν πολύ όπου ε, ότι η διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας ε, είναι πρόβλημα. Τέλος, ε, το παλιό σύστημα. Προφανώς λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που λειτουργεί εδώ και 100 χρόνια, οπότε η κληρονομιά του παλιού συστήματος είναι λογική να αναπτύσσεται με, μέσα στο εθνικό πλαίσιο και με κανόνες που είναι εθνικοί. Αυτό αντιμετωπίζεται. Ήδη το εξετάζει ο οργανισμός, το είπαν και σε κάποιες παρουσιάσεις, αλλά απαιτεί χρόνο μέσω των TSI και της δημιουργίας νέων υποδομών να υπάρξει εναρμόνιση. Παραμένουν βέβαια και μια σειρά εθνικών κανόνων που δημιουργούν ή στηρίζουν αυτά τα εμπόδια εισόδου. Για παράδειγμα υπάρχει έλλειψη διαφάνειας πολλών εθνικών κανόνων. Συχνά ο κατεστημένος έχει και πλεονέκτημα γνώσης σε σχέση με τον εισερχόμενο που δημιουργεί εμπόδιο, ενώ υπάρχουν και κάποιοι περιττοί εθνικοί κανόνες που ανέφεραν ορισμένοι εμπλεκόμενοι φορείς. Αν μπούμε τώρα λεπτομερέστερα στο μελλοντικό ρόλο της, ε, του, του, του οργανισμού. Ακούσαμε και το πρωί και, και τώρα ότι οι περισσότεροι συμφωνούν πως ο καλύτερος τρόπος μείωση ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο ο οργανισμός στην διαδικασία πιστοποίησης και διοδότησης για να περιοριστούν ο αντίκτυπος κάποιων προβλημάτων ή και για να εξαλειφθούν τελείως. Στην ανάλυση που κάναμε εξετάσαμε μια σε αναλλακτικών λύσεων. Από την προσέγγιση δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή το status quo, μέχρι μια προσέγγιση όπου τα πάντα τα κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και πάβουν να υφίστανται οι εθνικές αρχές. Και προφανώς υπάρχουν και διάμεσες ε, εναλλακτικές που δεν μπορείτε να τις δείτε καλά στην οθόνη. Η μαύρη γραμμή είναι η βασική γραμμή και που προχωράει σε μεγαλύτερο συντονισμό. Η άλλη περίπτωση είναι όταν ε, ο οργανισμός είναι one-stop shop, στην τρίτη όταν ε, η τελική απόφαση είναι του, ε, των εθνικών αρχών και στη κόκκινη γραμμή είναι όταν η τελική, το τελικό OK το δίνει η ο Ευρωπαϊκός Φορέας. Και βλέπετε ότι ανάλογα με το κόστος αδειοδότησης, ότι και στην τελευταία περίπτωση η φυστάμενη κατάσταση θα επιτρέψει βελτίωση στο, στη μείωση του κόστους αλλά οι άλλες εναλλακτικέ δίνουν μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, μεγαλύτερα κέρδη στον κλάδο. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος ε, πιστοποίησης ασφάλειας, όπου τα πλεονεκτήματα βελτιώνουν, αυξάνονται, τα, τα έσοδα αυξάνονται ανάλογα με τις επιλογές που κάνεις. Η ανάλυση ωστόσο συνολικά δεν στηρίζεται μόνο στους φορείς και τους κατασκευαστές. Εξετάζει και τον αντίκτυπο συνολικότερα στον κλάδο. Το κόστος για τον οργανισμό με τους νέους ρόλους ή το κόστος για τις εθνικές αρχές όταν παράγουν νέους ρόλους. Συνολικά λοιπόν η επιλογή που θεωρήσαμε καλύτερη είναι όταν ο οργανισμός μοιράζεται αρμοδιότητες με τις εθνικές αρχές ασφάλειας ότι την τελική απόφαση για την πιστοποίηση και την αδειότητα την παίρνει ο, οργανισμό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, αλλά χρησιμοποιεί όπου είναι αναγκαίο εθνικούς εμπειρογνώμονες των εθνικών αρχών. Μεσοπρόθεσμα θα χρειαστούν, βράχη πρόθεσμα θα χρειαστούν πολλοί τέτοιοι, ενώ όσο δηλαδή βελτιώνει την ε, γνώση της η, ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Διονόρη. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Επομένως τώρα οι τρεις συγητές, Μπιλμπάο, Κράμερ και Ζίλερ έχουν πέντε λεπτά ο καθένας και τρία λεπτά στη συνέχεια για τους ε, υπόλοιπους ε, συντονιστές και σε οποιοδήποτε άλλο μέλο επιθυμεί να πάρει το λόγο βέβαια. Πείτε μου το απλώς τώρα. Ξεκινάμε με την κυρία Μπιλμπάου για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με τις συζητήσεις το πρωί και τις συζητήσεις τώρα πιστεύω ότι έχουμε στα χέρια μας μια τεράστια πρόκληση και νομίζω και μια μεγάλη ευθύνη. Συμμερίζομαι πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν. Εγώ θα έκλεινα ωστόσο λέγοντας ότι υπάρχει κοινή διάγνωση για την ύπαρξη υπερβολικά πολλών κανόνων σε εθνικό επίπεδο, έλλειψη διαφάνειας των εθνικών αρχών, καθυστερήσει στην πιστοποίηση και την αδειοδότηση. Ωστόσο, η ανάγκη αλλά και η ανάγκη αλλαγή του status quo. Πιστεύω ότι με την έκθεση για την ε, διαλειτουργικότητα πρέπει, έχουμε την ευθύνη και πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση, μια προηγμένη ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί εν τέλει, έχοντας ακούσει ό,τι άκουσα, διαπιστώνω ότι οι ιστορικές επιχειρήσεις στις χώρες ε, που έχουμε ως αναφορά είναι αυτές που προσπαθούν να διαφυλάξουν το status quo. με συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και υπουργείων. Εδώ σε διάφορες εκθέσεις του Κοινοβουλίου είδαμε ότι εν γέννη οι εθνικές αρχές έχουν την τάση και ελπίζουμε να αλλάξει η θέση αυτή με το τέταρτο πακέτο, έχουν την τάση πάντω να θέλουν να κρατήσουν το status quo. Τα στοιχεία που μας δόθηκαν σήμερα δείχνουμε ότι αυτή η στάση δυσχεραίνει την καινοτομία, την ανάπτυξη της, της αγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκά επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς προκλήσεις, έλλειψη διαφάνειας, που εμποδίζει την ιδιωτική επένδυση και δυσχεραίνει την πρόσβαση στην αγορά και δυσχεραίνουμε τη θέση της ε, ανάπτυξης. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην έκθεση και να επεξεργαστούμε μία έκθεση που θα μας στοιχήσει πολύ δουλειά να το συμφωνήσουμε, αλλά που θα προσανατολίζεται ώστε να έχει σημαντικό ρόλο ο οργανισμός, να απλοποιηθούν οι τεχνικές απαιτήσει και να διευκρινιστεί ο ρόλος των εθνικών αρχών και με όλα αυτά που είπα θέλω να ρωτήσω τον κύριο ε, τον κύριο Κορτάθρα για την παρέμβασή του. Είπε κάποιος ότι καθυστερούν ε, χρόνια για κάποια βαγόνια άκουσα ότι καθυστέρησαν 7 χρόνια να πάρουν άδεια. Ποιος είναι ο μέσος όρος για την έκδοση των αδειών. Πόσο αυξάνει η καθυστέρηση αυτή το κόστος των προϊόντων και πόσο αυξάνει το κόστος του προϊόντος στον τελικό χρήστη, στον τελικό καταναλωτή. Στον... Γιατί κάποιο την καθυστερήσει την πληρώνει. Δεν είναι τζάπα η καθυστέρηση. Ούτε την πληρώνει μόνο ο παραγωγό ή ο κατασκευαστή. Εν τέλει ο πελάτη θα καταβάλει το κόστος αυτό και θα πρέπει να το περάσει στον άλλο πελάτη Για να προχωρήσουμε λοιπόν προς μια ευρωπαϊκή ανάπτυξη του σιδεδόμου με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, θα ήθελα να ρωτήσω τι τι κόστος έχει η καθυστέρηση και η μη απλοποίηση. Στην μείωση των διαδικασιών. Συμφωνώ με απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Διονόρη, ότι χρειάζεται όλες τις αποφάσεις να τις έχουμε σε, πληροφορία, σε υποστήριξη πληροφορική. Εμείς ό,τι έχουμε τώρα το έχουμε ε, στο χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα μηχανογραφημένο. Θα πρέπει αυτό να είναι έτοιμο για όλους τους ε, ανταγωνιστές τους, ώστε να μπορεί να το συμβουλευτεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Κύριε Κορτάφερ, θα ήθελα να μου δώσετε κάποια στοιχεία για το κόστος αυτό, ουσιαστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπιλμπάου. Προτού πάρει το λόγο ο κύριος Κράμερ, θα ήθελα να καλωσορίσω μια άλλη ομάδα επισκεπτών, επισκέπτες της κυρίας Γκέπχάρτα από την περιοχή της Στουτγκάρδης. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών και ελπίζω πραγματικά να βρείτε ενδιαφέρουσα τη συζήτηση αυτή. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Νομίζω η ανάλυση είναι σωστή. Το σύστημα στην Ευρώπη είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και δεν ε, εξυπηρετεί τους σιδηροδρόμους. Πρέπει να αλλάξει. Απογοητεύομαι όμως από πολλά κομμάτια των εκθέσεων που αναφέρουν τα άσχημα και γιατί είναι άσχημα. Τα ξέρουμε αυτά. Εγώ περίμενα συγκεκριμένα να πείτε εδώ έχει δίκιο η Κομισιόν, εδώ χρειάζονται βελτιώσεις και να έρθουν βελτιωτικές προτάσεις. Δεν άκουσα πολλά ε, άκουσα ότι η προβληματική RTM, TSM ε, ε, παρουσιάζεται ξανά και τώρα έχουμε το ίδιο σύστημα όπως και πριν. Διαφορετικά συστήματα πάνω στη βάση του ERTMS και αυτό πρέπει να το δούμε. Το μόνο είναι σωστό. Δεύτερον, η Ολλανδία η επιτάχυνση είναι σωστή, αλλά το unbundling είναι καταστροφικό, το είπαν κι άλλοι. Παρ' όλα αυτά ε, θέτω το ζήτημα. Με ή χωρίς unbundling υπάρχουν διακρίσεις. Ποια είναι η θέση σας εδώ και πώς εκτιμάτε το κόστος. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει πρόβλημα, θα κερδίσουμε λεφτά. Οι άλλοι λένε θα στοιχήσει 5 δις. Τι γίνεται ο καθηγητής από την Ισπανία και το TSI. Καλό είναι αυτό και όχι μόνο επειδή είναι εδώ η ομάδα της Τουτουγάρδη. Πρέπει να πω ότι στη Τουτουγάρδη κατασκευάζεται νέο σιδηροδρομικό σταθμό για 10 δι και νέε γραμμέ. Το σιδηροδρομικό σταθμό ε, είναι μικρότερε ικανότητε από το παλιό και αυξάνεται το κόστος στη μεγάλη και το 70% των επιβατών ε, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν εκεί αλλά έχει νόημα όπως και η γραμμή Παρίσι-Μπρατισλάβα όμως ε, θα πρέπει να δούμε ε, ε, το κόστος, ιδιαίτερα στους εμπορευματικούς σύρμους. Χρειάζεται συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές η διαφορά είναι μεγάλη και δεν ανταποκρίνεται στο TSI. Τι χρειάζεται το TSI εν τη αυτή περιπτώσει αν παραβιάζεται συνεχώς και όταν έχουμε συγχρηματοδότηση ε, επίσης δεν το καταλαβαίνω. Στις βαλτικές χώρες ήταν καλό αυτό που είπατε για τα μεμονωμένα δίκτυα, αλλά δεν είστε μεμονωμένο δίκτυο σε μια χώρα, Τέσσερι. Και ένα κομμάτι της Πολωνίας, Λιθουανία, Εσθονία, ε, Λετωνία και οι τέσσερις. Δεν μπορούμε να έχουμε εξαίρεση για ένα κράτος, αλλά για κάποιο σύστημα. Ή στην Ιβηρική, Πορτογαλία, Ισπανία. Εδώ τι θα κάνουμε βεβαίως, ε, υπάρχουν εθνικές ιδιαιτερότητες. Τελειώνω. Ε, δεν βλέπω τη νομική βάση στο νέο σύστημα για τον ΕΟΣ. Ε, ούτε η Κομισιόν μας το είπε. Τι καθήκοντα θα έχει. Και εκεί δεν είπε τίποτα η Κομισιόν. Χρειάζεται σαφή καταμερισμό εργασία. Δηλαδή αυτό θα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμω ε, τούτη και οι άλλοι τομεί ε, θα εμπίπτουν στου εθνικού φορεί. Αλλιώ θα γίνονται όλα δύο φορέ και δεν το θέλουμε. Οι εθνικοί φορεί λοιπόν που θα πρέπει να μειωθούν για να διαθέσουν ε, και να μεταθέσουν αρμοδιότητες στον ΕΟΣ. Ε, δεν μπορεί ο ΕΟΣ να τα αναλάβει όλα. Δεν μπορεί δηλαδή, θα πρέπει να προσλάβει 30.000 ανθρώπους. Δεν γίνεται, δεν πρόκειται περίπτωση. Αλλά το 95% ε, θα παραμείνει, νομίζω, σε εθνικό επίπεδο. Αλλά αν υπάρξει σύγκρουση και αν κάποιος πει όχι, ε, δεν θα δώσουμε άδεια σε αυτό το, σε αυτό το τρένο από την Γαλλία και θα πει ο ΕΟΣ όχι, η άδεια ισχύει για τα 25-26 κρατημέλη. Ποιο θα επιβληθεί τότε, ποιανού θα περάσει, ποιο θα έχει τον τελευταίο λόγο. Σε περίπτωση σύγκρουση θα πρέπει να είναι σαφέ λοιπόν ότι ο ΕΟΣ θα έχει τον τελευταίο λόγο για να ξέρουν όλοι ότι ε, γίνεται έλεγχος ε, ε, πριν αποφανθούν. Κάποιες, ε, κάποιες τεχνικές προδιαγραφές χρησιμοποιούνται για να υπάρξει η ανταγωνιστικότητα του δικτύου. Υπήρξαν κάποιες ε, ε, απάτες που αποκαλύφθηκαν, άλλες όχι. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες για τον ΕΟΣ που πρέπει να τα παρακολουθεί αυτά. Δεν υπάρχουν τώρα και πρέπει να διευκρινιστεί τι θα κάνει. Και ποιο είναι ας πούμε για εσάς η κόκκινη γραμμή για τις εθνικές αρμοδιότητες και πού θα πρέπει να παρεμβαίνει το Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Ο κύριος Σέλερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και όλους τους παρόντες συνεδρίαση αυτή, τους προσκεκλημένους μας, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και παρουσίαση που ακούσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία έχω συμπεριλάβει και εγώ στη δική μου την έκθεση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να συγκεράσουμε τα διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τόσο διαφορετικά. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ορισμένες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν εντελώς τα συστήματα, εθνικά συστήματα ασφάλειας, άλλες πάλι που τις χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές πολύ λιγότερο και αναφέρονται περισσότερο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντεροδρόμων. Βλέπουμε και το κόστος ότι κυμαίνεται από μηδενικό έως 10 εκατομμύρια. Αυτό ακούσαμε στην παρουσίαση. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε ένα καλό κοινό σύστημα το οποίο θα έχει την απαραίτητη ευελιξία και θα δίνει επιλογές για τους πελάτες, καθώς επίσης και για τις δρομικές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να επιβαρύνονται και να τιμωρούνται τελικά από ένα κοινό σύστημα το οποίο θα πρέπει να επιβληθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ιδανικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, κύριε Διονόρη, μπορείτε να μας πείτε ποιο θα είναι το λογικό κόστος όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αν μπορείτε να μου πείτε θα ποιο θα είναι το κόστος όσον αφορά την επαλήθευση της ασφάλειας, τον έλεγχο της ασφάλειας. Αγγίσουμε βέβαια σιγά σιγά και κάποια άλλα ζητήματα και νομίζω ότι από την οδηγία αυτή οι κατασκευαστέ είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφεληθούν περισσότερο. Από την άλλη υπάρχει μια κάποια σύγχυση και αυτό φάνηκε και συζητήσει που είχαμε με προσώπου του κλάδου και ενδιαφερομένους. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει γενικότερη βούληση να δοθεί περισσότερη αρμοδιότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων προκειμένου να αδειοδοτεί και τα εξαρτήματα θεωρείτε ότι ο κλάδος θα μπορούσε να δώσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων προκειμένου να τυποποιήσει τελικά το, τα διάφορα εξαρτήματα του, της σιδηροδρομικής υποδομής. Και να έλθω σε ένα ζήτημα τώρα το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα. Έχουμε πολλές διαφορετικές ε, καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία υπάρχει η δυνατότητα ρωσικούς σιδηροδρόμους να έρθουν στην ε, Φιλανδία, να κυκλοφορούν ελεύθερα και να φτάσουν στην Φιλανδία. Το αντίστροφο όμως δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τόσο ελεύθερη πρόσβαση για τα φιλανδικά τρένα προς την ε, Ρωσία. Στις υπόλοιπε βαλτικές χώρες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν κάποιο έχει καταγραφεί σε ένα μητρό που υπάρχει στη Μόσχα, νομίζω ότι μπορεί τότε τα τρένα της χώρας αυτής να κινηθούν πιο εύκολα προς τη χώρα αυτή και προς τις βαλτικές χώρες. Ουσιαστικά όμως αυτή τη στιγμή έχουμε μετακινήσεις περισσότερο από τις βαλτικές χώρες προς τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία και όχι τόσο προς υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δημιουργηθεί λοιπόν μία υπηρεσία, μία στάση στην Βαλένθια, ποιος τελικά θα επωφεληθεί. Θα επωφεληθούν και χώρες όπως η Φιλανδία ή οι βαλτικές χώρες ή θα διατηρήσουν τελικά τη βάση δεδομένων τους και το σύστημα πιστοποίηση στη Μόσχα. Και αν υπάρχει αυτή η υπηρεσία μια στάση στη Βαλένθια, τότε θα μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια και μοναδική ενιαία ευρωπαϊκή έγκριση για την υποδομή την οποία χρησιμοποιούμε και στις δικές μας περιοχές. Νομίζω πρέπει να δούμε τώρα ακριβώς πώς λειτουργούν και οι συνδρομικές επιχειρήσεις, ειδικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε μονομένε χώρες. νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε επιχειρήσεις αυτές και όχι τόσο στις δρομικές επιχειρήσεις των τρίτων χωρών. Όσον αφορά τα μεμονωμένα δίκτυα, ξέρετε ότι για τις μηχανέ είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε από την Εστονία στη Λετωνία. Ο Τόμας Χίρελ, πρώην συνάδελφό μα, πρόεδρος τώρα τη Εστονία, είχε θελήσει ουσιαστικά να έρθει εδώ πέρα χρησιμοποιώντας σιδηρόδρομο, τον υφιστάμενο σύστημα το οποίο υπάρχει δηλαδή στη χώρα του. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι η Εθνική Αρχή Ασφάλειας της χώρας του χρειάστηκε να κάνει πρώτα μία επαλήθευση για να δει τελικά αν θα μπορούσε να γίνει το ταξίδι αυτό και θα μπορούσε να γίνει αυτή η μετακίνηση. Και βρεθήκαμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης ε, των ε, πιστοποιήσεων ασφάλειας για τα μεμονωμένα δίκτυα, για όλες αυτές τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν μεμονωμένα δίκτυα. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση σε τρία στάδια για τη συνεργασία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και τι σε εθνικές αρχές ασφαλείας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ του ομιλητέ. Η Μπέλγα, το πρακτορείο ειδήσεων, σήμερα ε, ε παρουσία, λέει το εξή. Δεν μπορούν τα τρένα της SNCB να πάνε στο Λουξεμβούργο και έχω μείνει στην Αρλόν λόγω έλλειψης αδειοδότησης από τους... Και λέει ότι το Βέλγιο στον τομέα του ασφάλεια έχει κάνει συστηματικές επενδύσει. Και λέει. Η διοίκηση των συνδεδόμων του Λουξεμβούργου διαβεβαίωσε ότι του επόμενου μήνε το θέμα θα λυθεί. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, οι επιβάτε πρέπει να κατεβούν από το τρένο στο Αλόν και να ανέβουν σε άλλο τρένο για το Λουξεμβούργο. Αν θέλετε μια περίληψη, αυτό που θέλουμε εμεί να επιτύχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αυτό είναι να αποφευθεί ακριβώ αυτό που λένε από το Βελγικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γιατί μετά θα έρθουν και θα μας πούνε τι κάνετε εσείς στην Ευρώπη για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί λέτε ότι είναι οι οδικές μεταφορές αποτελεσματικές και οι σιδηροδρομικές όχι όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και ο προσανατολισμός είναι αυτός που ακούσατε. Εσείς πιστεύετε ότι οι τωρινές προτάσεις της Κομισιόν δίνουν άμεση σαφή απάντηση σε όλα αυτά αν ναι, πού και αν όχι, τι πρέπει να βελτιώσουμε εμείς οι βουλευτές για να επιτευχθούν οι στόχοι που βρίσκουν από ό,τι άκουσα σύμφωνους όλους. Αυτό είναι το πρώτο συγκεκριμένο ερώτημα. Δεύτερο, παρόμοιο με αυτό που είπε ο Μίχαελ, ο Μίχαελ Κράμερ πριν από λίγο, θέλω να μου πείτε για τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, γιατί δεν είναι σαφής πώς θα μοιραστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας και των Εθνικών Υφισταμένων Αρχών, γιατί πρέπει να υπάρξει μια μορφή συνεργασίας μεταξύ τους. Και ποιο θα είναι ο επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, ούτω ώστε αυτό ο νέο καταμερισμό να μην οδηγήσει σε γραφειοκρατικά και ε, τεχνολογικά εμπόδια. Πώς θα μπορέσουν να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος, ε, ερώτηση διευκρινιστική. Μιλήσαμε για την πιστοποίηση και τη διαδικασία. Ε, φτάσαμε σε 1,6 δις ευρώ που είναι τα περιουσικά στοιχεία που περιμένουν διοδότηση. Θέλω να καταλάβω ποιο είναι το γραφειοκρατικό κόστος εδώ και ποιο είναι το τεχνολογικό κόστος. Τι μπορούμε γρήγορα να το αντιμετωπίσουμε και πού πρέπει να επενδύσουμε στο ακόμα στο βαθμό που δεν υπάρχει τεχνολογική εναρμόνιση. Ευχαριστώ. Αλκαντράου, οι τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους ομιλητές για την παρουσίαση που μας έκανε. Μια διαπίστωση κάνω. Πολύ σημαντικέ φαίνεται ότι είναι οι διαφορές μεταξύ των αριθμών αρχών ασφάλειας. Σε τέτοιο βαθμό που αναρωτιέμαι κάποιες εθνικές αρχές μπορούν σήμερα να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Εγώ έχω αμφιβολίες. Με βάση τις πρώτες συζητήσει που έγιναν μεταξύ κρατών μελών στο περιθώριο του Συμβουλίου, θα έλεγα ότι τα κράτη προσπαθούν να καθυστερούσουν όσο μπορούν την υλοποίηση των ε, κανόνων ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο και στο μέλλον ακόμα εν τέλει, αυτή είναι η ερώτησή μου, θα μπορέσουμε αντί για αποπλοποίηση να... Υπάρχει κίνδυνος να επιδεινώσουμε, να περιπλέξουμε τα πράγματα, να τα απλοποιήσουμε. Να έχουμε δηλαδή πέραν του ευρω... του των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων να προσθέσουμε και ένα ευρωπαϊκό. Επαναλαμβάνω ότι η πρόοδος πρέπει να είναι πραγματική πρόοδος, όχι να πάμε πίσω. Και στο μέλλον το επίπεδο ασφάλειας θα πρέπει να είναι εξίσου υψηλό ή μη υψηλότερο από, αύριο από ό,τι σήμερα. Επ' αυτού θα κρυθούμε στο πακέτο αυτό και όλα θα εξαρτηθούν από την ποιότητα του Ευρωπαϊκού Συνδρομικού Οργανισμού. Και αμέσως το ερώτημα που τίθεται είναι πόροι, τεχνογνωσία, προθεσμίες, πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός αυτός σωστά. Οι συνάδελφοί μου το πανίδι, Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ενισχύεται, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ενισχύεται, ενώ οι εθνικές αποδυναμώνονται. Πώς θα διαμορφώσουμε την μετάβαση με σωστό τρόπο. Πώς θα είναι σαφές το πλαίσιο. Μακροπρόθεσμα ή μέσο πρόθεσμα θα πρέπει να ξέρουμε τι ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο και τι ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Αυτές είναι κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Κύριο Ντεμπάκη, ρίχνει το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την συμβολή τους, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα θέλω να θέσω. Ο εκπρόσωπος των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων, ΕΝΕΣ, μας είπε ότι υπήρχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την υποδομή και με κάποια άλλα επιμέρου στοιχεία των, της οδηγίας. Είπε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει αυτά να καθορίσουν πώς θα καθορίσουν τους στόχους, πώς θα επιτύχουν, με συγχωρείτε, τους στόχους που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί και πώς θα επαληθεύσουμε ότι έχουν όντως επιτευχθεί. Και τι θα γίνει σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν κάνει τίποτα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πώς θα καταφέρουμε να επιβάλλουμε στο κράτο μέλο αυτό μια πολιτική προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ξέρετε ότι αυτό που είδαμε στο παρελθόν είναι ότι θέταμε στόχου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάθε κράτος μέλος προσπαθούσε με τον δικό του τρόπο, ή πολλές φορές δεν προσπαθούσε, να πετύχει το στόχο αυτό. Μιλήσαμε επίσης για πολύ μεγάλες προθεσμίες. Είδαμε επίσης ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα ακόμα πολλές φορές και στο γειτονικές χώρες όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια έγκρισης και διοδότησης. Νομίζω ότι θα πρέπει τόσο οι Εθνικές Αρχές Ασφαλείας αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδροδρόμων να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό. Αλλά ποιο θα έχει την κύρια αρμοδιότητα. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο μπορεί να βρεθεί η λύση αυτή, γιατί αν υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο πολύ ειδικέ γνώσει στο συνδρομικό τομέα, τότε θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να διαβιβαστούν οι γνώσεις αυτές και επομένως κατ' επέκταση και αρμοδιότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντηροδρόμων. Κατάλαβα βέβαια τι είπανε όλοι οι μιλητές ως προς αυτό και θα το λάβω υπόψη μου στις μελλοντικές συζητήσεις που θα έχουμε. Ο κύριος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νιώθω σαν να βλέπω μια κακή ταινία. Όταν ε, ήταν ε, οδηγός σιδηροδρόμων ο παππούς μου, ταξίδευε σε όλη την Ευρώπη με το σιδηροδρόμο και δεν είχε τέτοια προβλήματα. Τώρα έχουμε προχωρήσει και έχουμε διαφορετική και προδιαγραφές για τον έλεγχο. Αν θέλουμε αποτελεσματική Ευρώπη στον τομέα των σιδηροδρόμων, αν θέλουμε έως αποτελεσματικό, γιατί να μην πάρουμε ένα πίνακα, να βάλουμε τις προϋποθέσεις όλων των, αργών, των αρχών πιστοποίησης για τους επιβάτες, ε, τα βαγόνια, την υποδομή, ε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τις απαιτήσει. Γιατί εδώ μπορεί να λέμε πολλά. Αλλά αν δεν μπορούμε στην πράξη να ενοποιήσουμε τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα, τους επιμέρους τεχνο, τεχνολογικούς εξοπλισμούς, όλοι θα γελάσουν μαζί μας. Παράλληλα, πρέπει να έχουμε συμφωνία άρσης πιστοποιητικών μεταξύ των ε, ε, αρχών πιστοποίησης. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι θα εξεταστεί, πώς, τι θα πιστοποιηθεί. Ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η συμφωνία. Χωρίς αυτή, όσο και να μιλάμε, δεν θα γίνει τίποτα. Ο συνάδελφος από, την, από το Πανεπιστήμιο λέει ότι υπάρχουν διάφορα, διάφορες δοκιμές που, πρέπει, που ε, αναφέρονται. Να τις δούμε. Να γίνουν από την αρχή ίδιες για όλους. Γιατί αν συνεχίζουμε να λέμε ότι έχουμε 17 διαφορετικές σειρές δοκιμών, τότε αυτό είναι τελείως λάθος. Δεν χρειάζεται επίση ένα ενιαίος οργανισμός, χρειάζονται ενοποιημένε διαδικασίες και αναγνώριση των πιστοποιητικών. Αν δεν το διασφαλίσουμε αυτό, τότε θα θεωρητικολογούμε και μόνο. Ευχαριστώ κύριε Κόλιτσεκ. Όταν ο παππούς σας ήταν σιδηροδρομικός, ήταν ε, ε, του ατμού η σιδηροδρομή που ήταν διαλειτουργική. Μήπως πρέπει να κάνουμε αυτό, να ξαναχρησιμοποιήσουμε τον ατμό, να πάμε πίσω στις ε, ατμομηχανές, δηλαδή πάλι στους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Στάνιεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πολλές συναντήσεις και νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση ότι χρειάζομαστε ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε ωστόσο τις διαφορές ε, των δικτύων με την ίδια μορφή ασφάλειας παραμένουν. Πρέπει να κοιτάξουμε το γιατί αυτό είναι δυνατό, όχι το γιατί δεν είναι δυνατό. Το πρωί μου ανέφεραν ε, τους λεγόμενους παντογράφους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν στα ηλεκτροδοτημένα δίκτυα της Βρετανίας για παράδειγμα, αλλά που μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσει παντογράφους που να λειτουργούν και στην Ευρώπη και στο Βρετανικό σύστημα. Άρα μπορούμε να βρούμε μια λύση που να έχει οικουμενικό χαρακτήρα και να είναι ένα πιστοποιητικό ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί να έχει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό που να ισχύει για αυτό και όχι για εκείνο το δίκτυο. Μου είπαν ότι στις βαλτικές χώρες υπάρχει κάτι διαφορετικό. Στη Σουηδία υπάρχει επίσης κάτι διαφορετικό. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, στην πράξη πώς θα το δούμε αυτό. Χρειαζόμαστε, είναι γεγονός, ένα ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Ποιος θα το εκδώσει, η ΕΡΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, οι Εθνικές Αρχές Ασφάλειας οι ίδιε θα το κάνουν, θα το δίνουν σε άλλους να το κάνουν. Πρέπει να το δούμε. Οι εξουσίες του ΕΡΑ σχετίζονται με τους σπόρους του ΕΡΑ. Χρειαζόμαστε μια εθνική, μια μεγάλη αρχή ή θα πρέπει κάθε εθνική αρχή να εκδίδει με βάση σύμβαση το πιστοποιητικό που μπορεί να το κάνει. Επίσης θέλω να ακούσω την απάντηση στα ερώτημα που έφεσε ο Μίχαελ για τις διαφορές, τις συγκρούσεις δηλαδή. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών που και αυτό θα έπρεπε να πάει στο αέρα κατά την άποψή μου. Κύριο Σαβάμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προσπαθήσω να μπω στο ίντερνετ και να καταφέρω να δω πώς λέγεται το, το, το, 22 στο IMBDA. Λέγεται εδώ πέρα ότι είναι μία παροδία μίας α, στρατιωτικής νοοτροπίας και μίας α, γραφειοκρατικής κοινωνίας. Θα αναφέρω αυτά για να πω το ακόλουθο. Μ' αρέσει αυτό το οποίο λέμε, βαθμιαία προσέγγιση και συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια αμοιβαία προσέγγιση, βαθμιαία προσέγγιση, με συγχωρείτε, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στηροδρόμων και τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας, προκειμένου να μην χάσουμε την εθνική εμπειρογνωμοσύνη. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Το άλλο εγχείρημα έχει ως στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, από όσο εγώ καταλαβαίνω τουλάχιστον. Αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε αυτή τη βαθμιαία προσέγγιση, νομίζω ότι θα καταναλώσουμε περισσότερο χρόνο και περισσότερα χρήματα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με του εαυτού μα και να ρωτηθούμε πραγματικά αν θέλουμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Συνεπώ, ο μόνος τρόπος που πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι τελικά να καταργήσουμε τις εθνικές αρχές ασφαλείας. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τότε ας εγκαταλείψουμε το όλο εγχείρημα, γιατί πραγματικά δεν θα καταλήξουμε σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε και χρειαζόμαστε στο εθνικό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα ή έχοντας παράλληλα μία ενιαία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπυροδρόμων. ξεκινήσουμε από αυτό και ας λύσουμε έπειτα στη συνέχεια με αυτή τη βάση τα υπόλοιπα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο πάλι στους εμπειρογνώμονές μας και να τους ζητήσω να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά με τη σειρά με την οποία πήραν το λόγο, έχοντας ο καθένας τρία λεπτά. Ο κύριος Γκορταζάρο Ο Ομπιέτα έχει πρώτο το λόγο. Μπορεί να απαντήσει παρακαλώ πολύ. να απαντήσω στην κυρία Μπιλμπάου. Ο μέσος χρόνος αδειοδότησης ξεπερνάει συχνά τα δύο χρόνια, που σημαίνει ότι έχουμε πολλούς μηχανικούς που δουλεύουν δύο χρόνια αντί να ασχολούνται με άλλα θέματα που μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα για τη χώρα, για την Ευρώπη και για τις επιχείρησεις κατά πάση πιθανότητα. Για το κόστος θα έλεγα ότι ποικίλει, αλλά είναι περίπου το 10% του κόστους του οχήματος, του, του βαγονιού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν επιπλέον και επιπλέον ε, κυρώσεις, επιπλέον ε, πρόστιμα όταν καθυστερεί. Υπάρχουν και καθυστερήσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες προβλημάτων. Προβλήματα που σχετίζονται με γραφειοκρατική διάσταση και κόσμος που ασχολείται με το να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις που σας είπα φτάνουν τα δύο χρόνια. Για άλλους που ρώτησαν τι θέλουμε να είναι το τέταρτο πακέτο. Τι κάνει το τέταρτο πακέτο. Το τέταρτο πακέτο μας παρουσιάζει τη νέα αέρα ως ένα μέλλον που πρέπει να το υποστηρίξουμε για να υπάρχει στην Ευρώπη μια ομοιογενής δουλειά μεταξύ όλων των χωρών. Να μπορούν όλοι να ξέρουν ποιες είναι οι απαιτήσει για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τρένο στη γραμμή, στις διάφορες γραμμές που ακολουθούν τα τρένα και το τέταρτο πακέτο, αυτό που δεν έχει είναι αρνητικά. Είπε ο κ. Κράμερ το πρωί ότι δεν είδε τίποτα το θετικό στι προτάσεις μα. Εγώ πιστεύω ότι η τωρινή πρόταση ω έχει περιλαμβάνει, έχει συζητηθεί, μιλήσαμε για τα προβλήματα και είπαμε ότι πιστεύουμε ότι η λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που είναι χρόνος και χρήμα, και να δουλεύουν οι δικοί μας σε πράγματα που μπορεί να κάνουν, που να μπορούν να κάνουν προς όφελος και της Ευρώπης. Τώρα, να τονίσω ότι είναι αναγκαίο οι εμπειρογνώμονες των εθνικών αρχών ασφάλειας να συνεχίσουν να δουλεύουν. Δεν μπορεί να χάσουμε την γνώση τους. Αυτή είναι η γνώση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η γνώση. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη γνώση που έχουν σε μια μεταβατική περίοδο δεν είναι δύο, τρία, πέντε χρόνια. Θα πρέπει να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση των ατόμων αυτών και να τους μετατρέψουμε σε κάτι που θα βοηθήσουν το μέλλον. Να ξέρουμε, να έχουμε στην Ευρώπη εμπειρογνώμονες που να ξέρουν τα θέματα τους και να έχουμε υπηρεσίες, δομές που θα μπορούν να στηριχθούν σε ανθρώπους που έχουν γνώση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει αυτός ο κόσμος είναι η μόνη διέξοδος για να είμαστε βέβαιοι ότι τα τρένα μας θα προχωρούν με την ασφάλεια που θέλουμε και θέλουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, Πρόεδρε. Ik, eh, ik wil even reageren op, eh, op de vraag die... Λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Ντεμπάκα. για την ε, Ολλανδική προσέγγιση στις παραχωρήσεις και ποιος πρέπει να είναι το μέλλον. Πρόκειται κυρίως για την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης. Πώς θα την ισχυροποιήσουμε τη θέση αυτή όσο μπορούμε. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ε, σε κάποιο επίπεδο, σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης και στην Ολλανδία. Εμείς θέλουμε να αυξηθεί ε, να αυξηθούν οι επιβατικές μεταφορές. Πώς θα γίνει αυτό. Στην Ολλανδία, αν δω τι θέλουν οι Ολλανδοί επιβάτες, θέλουν άμεσες συνδέσεις, ε, χωρίς μετεπιβίβαση και αν δούμε την υφιστάμενη κατάσταση λέμε ότι το 75% ε, θέλουν άμεση μεταφορά. Η μετεπιβίβαση μειώνει την ικανοποίηση των ε, επιβατών. Γι' αυτό θέλουμε το δίκτυο να ε, μην κατακαιρματιστεί, να λάβει υπόψη τις επιθυμίες των πελατών. Επίσης, ε, στο θέμα των παραχωρήσεων και οι επιχειρήσεις θέλουν να ικανοποιούν τον πελάτη, να υπάρχει ακρίβεια και τα παρόμοια. Αυτό θα συμβάλλει και στο μέλλον στην επιτυχία του πακέτου του, της τέταρτης δέσμης μέτρων. Ο κύριος Γκαρσία. Αναφέρθηκε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ εθνικών οργανισμών και ΕΟΣ, ο ΕΟΣ θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση. Αλήθεια είναι αυτό αλλά πρέπει να προσθέσω ότι μάλλον οι αρμοδιότητες του ΕΟΣ μετά τη λήψη απόφασης για την επίλυση κάποιας διαφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ποιος ελέγχει τον ελέγχοντα, ποιος ελέγχει λοιπόν τον φορέα ελέγχου και τι γίνει αν μετά από αυτή τη διαφορά η λύση που θα δώσει ο ΕΟΣ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων δηλαδή δεν είναι η ενδεδειγμένη. Κατόπιν τούτου δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το πρόσθετο κόστος. Αναφέρθηκε ήδη ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι ένα ε, επίπεδο πρόσθετων κανονισμών πέρα από τις εθνικές αρχές ασφάλειας που είναι το πρώτο επίπεδο και θα έχουμε και το δεύτερο επίπεδο, το πρόσθετο επίπεδο του ΕΟΣ. Και αυτό αλήθεια είναι, αλλά σε τελευταία ανάλυση κάποια πράγματα δεν θα αποτελέσουν πρόσθετο κόστος, γιατί πάντα γίνονταν έτσι. Επίσης αναφέρθηκε και το παρουσιάζω ως παράδειγμα ότι υπάρχουν 17 διαφορετικές δοκιμές. Αλλά αυτές δεν είναι διαφορετικές ε, για κάθε χώρα, απλώς είναι κάποια ανοιχτά ζητήματα. Και αν δείτε όλα τα TSI, τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, θα δείτε ότι συνεχώς ε, επικαλούνται χρήσιμα πρότυπα, τα οποία άλλωστε ήταν σε χρήση εδώ και δεκαετίες στον κλάδο των σιδηροδρόμων. Ε, δηλαδή υπενθυμίζουν το IUC ε, φυλάδιο ή τα πρότυπα τάδε. Αυτό δεν σημαίνει πρόσθετες εργασίες. Αντίθετα, καμιά φορά έτσι απλουστεύονται οι διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πέρης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι ένα σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και τη εργασία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στερεοδρόμου και των Εθνικών ε, Αρχών Ασφαλεία μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο μέλλον. Και αυτό δώσει και πολύ θετικέ λύσει για τα μονομένα δίκτυα. Όπω είπε ο κύριο Ζήλε, ο οποίος αναφέρθηκε στην χρήση μηχανών για διασυνοριακές μεταφορές ή για ταξίδια προς τρίτες χώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις αυτές απλή περιφερειακή μετακίνηση. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα που εντοπίζονται με σε όλες αυτές τις μεταφορές. Επίσης, Θεωρούμε ότι με το νέο αυτό σύστημα που προβλέπεται στον κανονισμό, στην οδηγία μάλλον, θα έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και μείωση του χρόνου που απαιτείται για, το, για την πιστοποίηση ασφαλείας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Και νομίζω ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, στα πλαίσια του οποίου θα ολοκληρώνεται μια διαδικασία πιστοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριος Διονόρη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αναφερθώ και εγώ σε κάποια σημεία όσον αφορά το μέσο χρόνο που απαιτείται. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο να σας δώσω ένα συγκεκριμένο αριθμό αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. Στη δική μου παρουσίαση αναφέρθηκα σε απόκληση πολλών ετών. Αλλά πάντως έχουμε, για παράδειγμα, αδειδότηση μηχανών σε τρεις μήνες, μέχρι αδειοδότηση η οποία μπορεί να πετήσει τρία χρόνια ή πολλές φορές και εφτά χρόνια για κάποιες αμαξοστοιχίες, οι οποίες σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να πετούν μόνο τρεις μήνες. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω ένα μέσο χρόνο και ούτε θα εξυπηρετούσε τίποτα αυτό. Έχει να κάνει με το είδος του οχήματο, ο απαιτούμενος χρόνος, αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι εξαρτάται και από το αν πρόκειται για πρώτη αδειοδότηση ή για μια επαναδιοδότηση. Επομένως, να σας δώσω αυτή τη στιγμή έναν αριθμό θα ήταν κάπως αυθαίρετο. Κύριε Ζήλε, το ότι είναι λογική αδειοδότηση, ποιο είναι λογικό κόστο για την αδειοδότηση και για την πιστοποίηση και ποιο είναι λογικό εύλογο χρόνο. Προτού πάλι σα δώσω ένα αριθμό, πρέπει να σα πω ότι είναι λογική διαδικασία. Λογική διαδικασία είναι μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία που θα δημιουργεί την απαραίτητη νομική ασφάλεια που χρειάζονται και οι κατασκευαστέ αλλά και οι σιδεροδρομικέ επιχειρήσει, προκειμένου να καταφέρουν να έχουν και την πιστοποίηση ασφαλεία, αλλά μπορούν να κάνουν και τι απαραίτητε επενδύσει για να αδειοδοτηθούν τα οχήματά του εξασφαλιστεί αυτό, τότε μπορούμε να μιλήσουμε και για εύλογο κόστος. Πρώτα όμως θα πρέπει να τυποποιηθεί η ευρωπαϊκά διαδικασία και νομίζω ότι αυτό πήγε ο κύριος Κράμερ λίγο νωρίτερα. Και νομίζω ότι το, το παράδειγμα του κύριου Γκρόσιου όσον αφορά τα βελγικά τρένα που πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο είναι πραγματικά ενδεικτικό των προβλημάτων που έχουμε. Ο κύριος Γκρόσα έπειτα μίλησε στη διάκριση των αρμοδιοτήτων. Δεν είναι πολύ εύκολο να καταφέρουμε να κάνουμε μια απόλυτη διάκριση σε μια σύντομη συζήτηση όπως αυτή που έχουμε τώρα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί πάλι μια ασφάλεια για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους κατασκευαστές, ότι δηλαδή υπάρχει ένας φορέας, εμπροκειμένο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος μπορεί να πάρει τελική απόφαση βασιζόμενος σε ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες που μπορεί να έρχονται από εθνικό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι η έγκριση θα δοθεί αυτόματα. Πάντω, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντεροδρόμων αυτή τη στιγμή δεν έχει απαραίτητα όλη την εμπειρογνωμοσύνη από κάθε κράτο μέλο. Γι' αυτό το λόγο βασίζεται ακόμα στην εθνική εμπειρογνωμοσύνη. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντεροδρόμων μπορεί να δώσει, να αρνηθεί μια έγκριση, αλλά σε, μια, σε ένα μεταβατικό στάδιο πρέπει να εξαρτάται ακόμα και από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Και γι' αυτό βασίζεται ακόμα σε εθνικές αρχές ασφαλείας οι οποίε ε, παρέχουν αυτή την εθνική εμπειρογνωμοσύνη. Νομίζω ότι μακρηγόρησα όμως. Μία τελευταία παρατήρηση με την αδειά σα, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να διατηρήσουμε την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και ποιο ήταν ο ρόλο που θα πρέπει να δραματίσει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και ποιο ήταν ο ρόλο του οργανισμού αυτού στην ε, επίλυση ε, νομικών διαφορών. Ο οργανισμός ο οποίος έχει πάρει μια απόφαση, μπορεί να προσφεύγει και στην απόφαση αυτή, να γίνεται προσφυγή μάλλον στον οργανισμό αυτό για την απόφαση αυτή. Να υπάρχει δηλαδή ένας διαμεσολαβητής ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει την επίλυση των νομικών αντιπαραθέσεων. Θεωρήσαμε ότι δεν θα εμφανίζονται βέβαια τις αντιπαραθέσεις σε καθημερινό επίπεδο και ότι θα είναι πιο εύκολο να λυθούν τελικά. Κυρία Μπιλμπάου, έχετε ακόμα μία ερώτηση σύντομη, σας παρακαλώ. Βέβαια. Για τον κύριο Γκαρθία. Κάποιος ρώτησε ποιος ελέγχει την, τον οργανισμό και ποια είναι η λύση. Τώρα ακούσαμε μόνο τη θέση για ένα νέο χαρακτηριστικό. Τι προτείνετε. Δεύτερον, στην πρώτη παρέμβαση σας μιλήσατε για το πρόγραμμα Safe to Rail με πέντε γραμμές έρευνας. Πιστεύετε ότι το Πανεπιστήμιο με την έρευνα η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να συμβάλλει στην προβληματική που αναφέρουμε για το τέταρτο συνδρομικό πακέτο και τι μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ για τις δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ποιος ελέγχει τον οργανισμό. Αυτό είναι ένα θέμα που συχνά θέτουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Υπάρχει δηλαδή ένας οργανισμός που ελέγχει εθνικές αρχές και που κάποιος ε, κάνει μια αίτηση για να γίνει η μελέτη σε επίπεδο δικαιοσύνη, σε επίπεδο δικαστικό. Συχνά οι συγκρούσεις αυτές δημιουργούν αποφάσεις που δεν στηρίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά σε άλλα. Ενώ κανονικά οι αποφάσεις πρέπει να τηρούν, να σέβονται τεχνικά κριτήρια, αποκλειστικά τεχνικά κριτήρια. Συχνά, ωστόσο, άλλοι διαφορετικοί λόγοι ακούγονται για την ε, πρότασή σας έρευνας Safe to Rail. Μπορώ να σας δώσω το παράδειγμα αυτό για να το καταλάβετε. Οι, επιχειρη... οι κατασκευαστές μας εξηγείται μάλλον ότι οι διαδικασίες ε, έγκρισης τύπου είναι μακρές και απαιτούν χιλιόμετρα δοκιμών, την παρουσία του οχήματος ε, στις γραμμές για μέρες και μέρες, χωρίς ε, χωρίς κέρδη. Δηλαδή είναι το, το τρένο εκεί πηγαίνω έχετε χωρίς να τόνι σιδήρου και χάλιβα που δεν, ε, που δεν δίνουν αποτελέσματα. Η σύγχρονη εξέλιξη επιτρέπει προσωμιώσεις που έχουν ακριβώς την ίδια, το ίδιο αποτέλεσμα και που σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε προσωμιώσεις για να κάνουμε τις ε, δοκιμές αυτές χωρίς το τρένο να κινείται φυσικά. Κάτι που θα είναι θετικό και για την επιχείρηση, για το τρένο και τους πολίτες. Ένα ε, ερευνητικό πρόγραμμα όπως αυτό το Safe to Rail στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 μπορεί να αυξήσει τη γνώση και να οδηγήσει σε βελτιώσεις που θα μειώσουν το κόστος και θα επιτρέπει τα τρένα να είναι σε καλύτερη υπηρεσία και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί παντού η ασφάλεια πρέχει. Τελειώσαμε με, με μακρά συζήτηση, ενώ νομίζω θα, θα τα είχαμε κλείσει πα, γρήγορα γρήγορα. Η Επιτροπή έχει είχε μιλήσει τρία λεπτά το πρωί ε, ούτε τρία λεπτά δεν είχε μιλήσει. Αν καταφέρετε να τηρήσετε το τρίλεπτο. Ευχαριστώ που μου δώσατε και το λόγο το πρωί. Φτάνουν τα τρία λεπτά. Καταρχήν ευχαριστώ για την ακροάση. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή και τους συζητητές για την ε, ωραία αυτή εκκίνηση στην εξέταση της τέταρτης δέσμης που είναι ολοκληρωμένη και θέλει να ολοκληρώσει τον ενιαίο σιδηροδρομικό ευρωπαϊκό χώρο. Τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του πακέτου της τέταρτης δέσμης είναι η ενιαία διοδότηση και σημαντικός ρόλος κεντρικός για τον ΕΟΣ που είναι ανεξάρτητος διαχειριστής υποδομών ε, και παρακολούθησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των κατεστημένων και βέβαια θα, με όλα αυτά θα επιτύχουμε τον ενίο σιδηροδρομικό χώρο. Χαίρομαι που αρχίζει λοιπόν τόσο γρήγορα η δουλειά στην Επιτροπή Μεταφορών. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα σχετικά με το τι είναι το η τέταρτη δέσμη μέτρων αφορά τους σιδηροδρόμους ως σημαντικός τρόπος μεταφοράς που πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο στα πλαίσια ε, ενός συστήματος βιώσιμου ενοποιημένου, ολοκληρωμένου. Προφανώς υπάρχει και φιλοδοξία του κλάδου, συζητήθηκε εδώ και χαίρομαι που μιλήσαμε για την πρωτοβουλία αυτή του κλάδου, το Shift to Rail, που συμπληρώνει κατά πολύ το τεχνικό πυλώνα του εις τέταρτης δέσμης μέτρων σε μια πλήρη εσωτερική αγορά ναι, και όχι με 25 διαφορετικά εθνικά συστήματα θα μπορέσει να αναπτύξει ο σιδηροδρομικός κλάδος προϊόντα που θα πουλήσει στην Ευρώπη, που θα τα λειτουργήσει αποτελεσματικά στην Ευρώπη και που θα πολλούνται και διεθνώς ε, με ε, ε, ανταγωνιστική, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κοινωνική διάσταση εδώ είναι σημαντική επίσης, αφορά την απασχόληση, συνθήκες απασχόλησης και υπάρχουν θέματα με τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που τα γνωρίζουμε και πρέπει να τα καταπιαστούμε και πολλά στοιχεία του, της δέσμης Ιδιαίτερα η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ε, ε, παρέμβει αν ε, αλλάξει μετά το διαγωνισμό ο ανάδοχος ε, είναι ένα θέμα. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους χρήστες, τους πολίτες που χρησιμοποιούν σιδηροδρομικές υπηρεσίες για να πάνε το πρωί στη δουλειά τους και να γυρίσουν το απόγευμα και την τέταρτη δέσμη μέτρων θέλει να διασφαλίσει ότι οι σιδηρόδρομοι θα μπορέσουν να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες και μετά βέβαια οικονομική διάσταση με την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικό σύστημα σιδηροδρόμων για την οικονομική μας ανταγωνιστικότητα. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και το κόστος. Η τέταρτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές θα βοηθήσει να μειωθεί το κόστος του σιδηροδρόμους. Ήδη αναφέρθηκε αυτό το θέμα το απόγευμα όταν μιλήσαμε για το τροχαίο υλικό. Αυτό ισχύει και για τα κόστη για το δημόσιο όταν μιλάμε για ε, αποζημιώσεις αντισταθμίσεις για υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και το κλάδος δουλεύει, τα κράτη-μέλη δουλεύουν, εμείς επίσης, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μειωθεί το κόστος του σιδηροδρόμου και ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να γίνει αυτό έχει δοκιμαστεί ήδη σε κάποια κράτη-μέλη και είναι η διαγωνιστική διαδικασία. Και αν το δούμε στην ε, μελέτη επιπτώσεων, και αν δούμε και τις εμπειρίες σε πολλά κράτη-μέλη, οι διαγωνισμοί στις δημόσιες ε, συμβάσεις μειώνει το κόστος ε, από 20 μέχρι και 30% καμιά φορά. Και τώρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη ως πολύ σημαντική πτυχή. Ξέρω ότι εξετάζεται από τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές. Αυτά σχετικά με το γενικό πλαίσιο για την παρουσίαση της τέταρτης δέσμης. Ε, τώρα κάποια επιμέρους σχόλια για τον τεχνικό πυλώνα που συζητήθηκε ε, πάρα πολύ ωραία σήμερα το απόγευμα. Εδώ επιβεβαιώνω και εγώ αυτά που συζητήθηκαν και ελέγχθησαν από τα μέλη της Επιτροπής αλλά και τους ομιλητές ότι το πακέτο στον τεχνικό πυλώνα, η τέταρτη δέσμη μέτρων δηλαδή, τι κάνει ε, κάνουμε το τελευταίο μίλη για την ολοκλήρωση ε, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας στους σιδηροδρόμου. Πολλά έγιναν τώρα από τη νέα νομοθεσία. Ο Μίχαελ νομίζω το είπε με πολλά παραδείγματα. Δεν καλύψαμε όλες τις εκκρεμότητες. Χρειαζόμαστε μόνο απευθυντική υπηρεσία και ενιαία διαδικασία με βάση αυτά που υπάρχουν τώρα όπου ο ΕΟΣ θα είναι ο βασικός ε, φορέας. Αυτό θα πρέπει να συνάδει και με τις εθνικές αρχές ασφάλειας, τις υπάρχουσες δομές ε, και δεν μπορούμε ε, ε, να φτιάξουμε ένα νεός που θα αντικαθιστά τις εθνικές αρχές ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να οργανωθεί σωστά η σχέση μεταξύ του ΕΟΣ και των Εθνικών Αρχών Ασφαλείας. Πρέπει επίσης να μειώσουμε απόλυτα τον αριθμό των εθνικών κανόνων. Αυτό είναι το προφανέστερο εμπόδιο για ολοκληρωμένους σιδηροδρόμους στην ενιαία αγορά. Ε, πολύ είναι ιστορικής ε, σημασίας που και δεν χρειάζονται πια. Ήδη ε, έχει αρχίσει η συζήτηση αυτή με τις εθνικές αρχές και γίνονται πολλά περισσότερα από όσα ξέρουμε, αλλά αυτά δεν αρκούν και η τέταρτη δέσμη μέτρων υποθέτει επίσης ότι αυτή η διαδικασία εξυγχρονισμού των εθνικών κανόνων θα ολοκληρωθεί, ούτως ώστε οι αδειοδοτήσεις να χορηγούνται μόνο πάνω στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν εθνικοί κανόνες, τα δίκτυα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη όταν ε, ε, λειτουργεί το τροχαίο υλικό με την αδειοδότηση που θα είναι ευρωπαϊκή και θα χορηγεί ε, με μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία. Τέλος, Ίσως αυτό δεν συζητήθηκε τόσο πολύ σήμερα το απόγευμα, αλλά δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της πρότασης, είναι ο σωστός επιμερισμός των ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΟΣ και Εθνικών Αρχών Ασφαλείας, το είπαμε αυτό, αλλά και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους τους σημαντικούς. Του φορεί ανάθεση, φορείς κοινοποίηση, ε, του διαχειριστέ, ε, των υποδομών, τι υδροδρομικές επιχειρήσει κλπ. Και θέλουμε να διευκρινίσουμε στην αναδιατύπωση τη οδηγία ε, για την ασφάλεια του αντίστοιχου ρόλου των κέριων, των κρίσιμων αυτών εμπλεκομένων, ούτω ώστε να γίνεται η διαχείριση τη ασφάλεια με πιο αποτελεσματικό τρόπο, αναθέτοντα τι ευθύνε εκεί που πρέπει. Και κάτι που δεν συζητείται πολύ είναι και η ευθύνη του κλάδου του ίδιου. Ε, βεβαίως το τεχνικό πακέτο ε, σκοπό έχει να βοηθήσει τους κατασκευαστές να έχουν ένα καλύτερο πλαίσιο εξυγχρονισμένο, καλύτερες ε, ταχύτερες αδειοδοτήσεις, αλλά διευκρινίζοντας τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του καθενός, ε, αυτό σημαίνει ότι θα φέρουμε αντιμέτωπο τον κλάδο με τις ευθύνες τους, γιατί κάποιες καθυστερήσεις πρέπει να αποδοθούν στον ίδιο τον κλάδο. Ε, χρειάζεται λοιπόν ένα καλύτερο, διαφανέστερο πλαίσιο και από αυτό θα ωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δύο σχόλια κύριε Πρόεδρε σχετικά με τη διακυβέρνηση. Θέλω να σας πω, κρίνοντας από τη σημερινή συζήτηση του πρωινού, ότι ο βασικός σκοπός της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι το unbundling, ο διαχωρισμός δηλαδή ιδιοκτησίας εκμετάλλευσης, αλλά ε, η θέσπιση ενός πλαισίου όπου οι διαχειριστές υποδομών θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης υποδομών και έτσι θα μπορούν να αναπτύσσουν εθνική υποδομή, θα αναπτύσσουν την υποδομή σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για να εξυπηρετούν όλους τους χρήστες των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι το πακέτο της διακυβέρνησης και εξετάζει τη σχέση με όλους τους παίκτες στην αγορά προτείνει επίσης Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Υποδομών για να υπάρχει σωστό πλαίσιο παροχών υπηρεσιών και επίσης καλύπτει και τη σχέση μεταξύ διαχειριστή ε, υποδομών και των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης και σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να πω ότι αν η πρόταση της Κομισιόν κάνει κάποιες προβλέψεις για να οργανώσει τη σχέση και να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της, είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί, ούτω ώστε οι προτάσεις να είναι αποτελεσματικές και σε σχέση με το κόστος και θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε εξυγχρονισμό των κανόνων διαχείρισης για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Έχουμε λοιπόν ε, εξυγχρονισμένο πλαίσιο, πλαίσιο ε, κοινή λογικής που διασφαλίζει την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομών. Τέλος, ε, μου είπαν για τα σχόλια σήμερα το πρωί ότι το unbundling δεν είναι μια πανάκια. Προφανώς αυτό είναι αλήθεια, αλλά ε, ούτε οι ρυθμίσεις ε, είναι πανάκια. Και αν δω τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές με κάποιες εξαιρέσεις, όλοι πιστεύουν ότι έχουν κεντρικό ρόλο να παίξουν και η αναδιατύπωση τους τον παρέχει τον κεντρικό αυτό ρόλο και τους σπόρους για να παίξουν το ρόλο τους, αλλά ε, πρέπει και οι διαχειριστές υποδομών να έχουν διαφάνεια και ανεξαρτησία από όλους τους εμπλεκομένους. Το, η τέταρτη δέσμη μέτρων, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, προσπαθεί να προσανατολιστεί στο μέλλον και να δώσει ένα πλαίσιο καινοτομία στους σιδηροδρόμους και είμαι βέβαιος ότι ο κλάδος θα ανταποκριθεί και γνωρίζω και ο συνομοθέτης θα ανταποκριθεί στο ρόλο του και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κύριε Πακέ. Για να κλείσω κι εγώ ως προεδρεύων. Ένα πράγμα που προκύπτει από την σημερινή συζήτηση είναι ότι όλοι ελπίζουν να μην υπάρξει πέμπτο πακέτο συνδρομικών ε, μεταφορών. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος. Τα θαύματα καθυστερούν. Αλλά φαίνεται ότι δείχνει την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όταν συζητούμε με τα σιδηροδρομικά θέματα. Ότι οτιδήποτε και θες να κάνεις με τα τρένα είναι πρόβλημα. Μου θύμισαν ότι πριν από 44 χρόνια ο άνθρωπος πάτησε την σελήνη. Ωστόσο, 44 χρόνια μετά την πρώτη προσελήνωση δεν μπορεί ένα τρένο από το Βέλγιο να πάει στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι τι άλλο να πω. Βλέπετε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Συχνά χρησιμοποιώ σαν αναλογία τις αερομεταφορές. Αν είχαμε τους ίδιους κανόνες ε, στις αερομεταφορές όπως αυτές που έχουμε στους ιδεοδρόμους ούτε ένα Airbus δεν θα, θα μπορούσε να πετάξει, διότι θα έπρεπε να πάρει 27 πιστοποιήσεις για το Α, 27 πιστοποιήσεις για το Β κτλ. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε ενοποίηση στις αερομεταφορές, γιατί να μην το κάνουμε στα τρένα. Και πρέπει να αποδεχθούμε ότι στο παρελθόν υπήρχε αυτή η τάση προστασίας των κατεστημένων επιχειρήσεων. Και το πρόβλημα είναι ότι τα τρένα δεν σκέφτονται πανευρωπαϊκά, ενώ τα αεροπλάνα σκέφτονται, έχουν ευρύτερο πλαίσιο. Οι ισιοδομικές επιχειρήσεις δεν σκέφτονται την διάσταση της Ευρώπης. Δεν σκέφτονται σχεδόν τίποτα πέραν των εθνικών ορίων. Μέχρι του αλλάξει η νοοτροπία, πάντα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Μπορείς να στείλει από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στο Χονγκ Κόνγκ ένα εμπόρευμα σε 13 ώρες, αλλά δεν μπορείς να στείλει τον ίδιο χρόνο ένα εμπόρευμα με τρένο από τη Μασσαλία στο Τράφοντ Πάρκ. Άρα δεν, δεν είναι λογικό. Κάποιοι συνάδελφοι το έθεσαν το θέμα του ρόλου της ΕΡΑ και στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο κανονισμός, ο Μάικλ το λέει αυτό συχνά στον κανονισμό TSI, κάπου κάπου αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχουν TSI, αλλά τα κράτη-μέλη δεν τηρούν την νομοθεσία της Ένωσης για τα TSI. Και η Αγγλία και η Βρετανία είναι μεταξύ αυτών, λένε. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι το βασικό θέμα δεν είναι ο διαχωρισμός. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι ο διαχωρισμός είναι σημαντικός. Κατ' εμέ ωστόσο, μέχρι ότου υπάρχει διαλειτουργικότητα, μέχρι ότου υπάρξει τεχνική εναρμόνιση που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα, δεν, τα υπόλοιπα δεν έχουν νόημα διότι και πάλι θα ζει σε ένα πλαίσιο όπου ο καθένας είναι στο εθνικό του σύνοράκι και θα κάνει την εθνική του δουλίτσα. Όντως, καταλαβαίνω την αντιμετώπιση με χωριστό τρόπο των ε, ε, απομονωμένων δικτύων. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα παλιά παραδοσιακά τρένα, τα, hate το heritage, το heritage goals, τις μικρές γραμμές. Αλλά αυτά είναι περιθωριακά θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω ωστόσο τους ομιλητές και από το απόγευμα και από το πρωί, τους συναδέλφους που ήταν παρόντες και όλους όσοι ήρθαν να ακούσουν την ακρόαση αυτή που ελπίζω ότι την βρήκαν χρήσιμη και ενημερωτική. Μην υποτιμούμε τη δουλειά που έχουν τώρα οι συνάδελφοι. Ακούσαμε τις αποκλίνουσες απόψεις. Ακούσαμε το ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο και είναι δύσκολο να μπορέσουν οι συγγητές να συνδέσουν τα πράγματα σε ένα κείμενο και να πείσουν τα μέλη της Επιτροπής μας ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Κατόπιν βέβαια έχετε δύσκολη για να πιστεί ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στους εισηγητές. Ξέρω ότι όλοι θα έρθετε για τις συζητήσεις, για τις τοπολογίες και τις εκθέσεις. Σας ευχαριστώ όλους. Κάποια οργανωτικά. Την Τετάρτη 29 Μαΐου η επόμενη συνάντηση 9 η ώρα. Σας ευχαριστώ όλους, Ευχαριστώ τους Γερμηνείς ο Πρόεδρος. Τέλος συνεδρίασης.